Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ για να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Please be seated. I would like to give a very warm welcome. Να καλωσορίσω θερμότατα την αυτοεξοχότητα των Σεήχη Μοχάμετ Μπίν Αμπτουλαρμάν Μπιντζάμιν Αλτάγιν, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό εξωτερικών του Κατάρ. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που βρίσκεστε εδώ στην Επιτροπή μας. Έχετε ξανάρθει βεβαίως. Θυμόμαστε ότι είχαμε μια εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων ε, και χθε το ε, απόγευμα, εγώ και εσείς. Όπως γνωρίζετε, οι τελευταίε εξελίξεις στην περιοχή του κόλπου είναι πολύ ανησυχητικές, ιδίω στο πλαίσιο των ε, αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Περισσότερο από ποτέ υπάρχει ε, επίγουσα ανάγκη αποκλιμάκωσης για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και παγκοσμίω. Εξοχότατε, θα θέλαμε να μα πείτε τι απόψει σα σχετικά με την κατάσταση τη εξελισσόμενη κρίση μεταξύ τη χώρα σα και άλλων χώρων εταίρων στην GCC. Γνωρίζουμε τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει το εμπάργκο εις βάρος του Κατάρ. Από την αρχή της κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν τηρήσει στάση ουδετερότητας και υποστηρίζουμε διαμεσολάβηση του Κουβέιτ στην επίλυση της κρίσης. Να υπογραμμίσω επίσης ότι η συνοχή ε, του Συμβουλίου Συνεργασίας των Αραβικών Χωρών του Κόλπου είναι κρίσιμη σημασίας για την υποστήριξη της περιφερειακής συνεργασίας σταθερότητας. Γιατί αυτή η κρίση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή και ευρύτερα. Τελικά, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων μεταξύ Κατάρ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και στον τομέα της ασφάλειας, στον τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων, της ενέργειας. Μας τα είπατε και χθε αυτά, αλλά ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε και ιδίω κάποιες περισσότερες πληροφορίε, ε, έπειτα και από την, συνεργασία, την συμφωνία συνεργασίας που υπογράφει, υπεγράφει σχεδόν πριν από δύο χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ να καλωσορίσω και τον πρέσβη σα, ο οποίο έχει μεγάλη δραστηριότητα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπετε ότι έχουμε και μεγάλη συμμετοχή ε, μελών τη της Έχουμε μαζί μα και τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Ήτρε και που μόλι είδα. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε για την πολύ ευγενική σας εισαγωγή. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχόμαστε επιτυχή θητεία. Επιτρέψτε μου να κάνω μια εισήγηση και μετά θα ακούσω βεβαίως ερωτήσεις και παρατηρήσεις σα. Είμαι εδώ στι για να ανταλλάξουμε απόψεις για να προχωρήσουμε στην εταιρική μας σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν της συνεργασίας σε περιφερειακά θέματα, θα γνωρίζετε ότι είμαστε μια μικρή χώρα σε μια ταραχώδη περιοχή και εντούτοι σε μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο. Διεθνώς υπολογίζουν σε εμάς για να διευκολύνουμε τον διάλογο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ίσως να μην γνωρίζετε ότι το Κατάρ υλοποιεί προοδευτικές εσωτερικές μεταρρυθμίσεις εδώ και δεκαετίες στα θέματα παιδείας, μετακινήσεων, αθλητισμού. Πλέον φιλοξενούμε πάρα πολλά δυτικά πανεπιστήμια στην Τόχα. Έχουμε προχωρήσει και στην ίδρυση του δικτύου Al Jazeera για ένα άνευ προηγουμένο επίπεδο ενημέρωσης. Έχουμε μία από τις καλύτερες εταιρείες αερομεταφορέων στον κόσμο και θα φιλοξενήσουμε βεβαίως και το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου το 2022 στην δική μας περιοχή και σας περιμένουμε. Ο πιο σημαντικός στόχος ανάπτυξης είναι να αντιμετωπίσουμε την εγκατάλειψη του σχολείου από τους μαθητές ε, και τον εναγκαλισμό τους από επικίνδυνες ιδεολογίες. Σε συνεργασία λοιπόν με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε επαναφέρει στο σχολείο 11 εκατομμύρια μαθητές και δημιουργούμε θέσεις, ε, ευκαιρίες για θέσεις απασχόλησης για 5 εκατομμύρια νέους ανθρώπους προάγουμε την ειρήνευση και την ευημερία σε όλη την περιοχή σε συνεργασία μαζί σας. Θεωρούμε ότι ο κόσμος, ο πλανήτης είναι συνδεδεμένος και οποιαδήποτε επιτυχία ή αποτυχία επηρεάζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και το αντίστροφο. Αυτή η διασυνδεσιμότητα προϋποθέτει συνεχή συνεργασία και προϋποθέτει πολυμερείς προσεγγίσεις και λύσεις. Στην περιοχή μας η πρώτη, η υπαριθμόν ένα πρόκληση είναι η ειρήνη και η σταθερότητα που θα επιτευχθεί μόνον όταν όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής, της περιοχής, βρουν συνένεση επί των πιο σημαντικών ζητημάτων. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία για όλους μας, διότι η σημερινή τρικυμιώδης, ταραχώδης κατάσταση έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες και για εμάς και για εσάς χρειάζεται μια συμφωνία ασφαλείας που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις χώρες της περιοχής ώστε να είναι βιώσιμη. Εμείς καλούμε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής να προχωρήσουμε σε δεσμευτικές ειρηνευτικές συμφωνίες και για να έχουμε τέτοιες συμφωνίες πρέπει αυτές να είναι συλλογικές επί τη βάση κοινών αρχών ειρήνευσης, λογοδοσίας, σεβασμού της κυριαρχίας των μελών και κοινή δέσμευση σε μη ε, επιρροή στα εσωτερικά θέματα εταίρων. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη τη διπλωματική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε κάθε χώρα της Μέσης Ανατολής να προσέλθει στο τραπέζι για να αποκαταστήσουμε την παγκόσμια τάξη της ειρήνης. Θα αποκλιμακώσουμε τις ε, συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Πρόσφατα είχαμε και καλά νέα στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ταλιμπάν που φιλοξενούμε στην Τόχα. Αυτό είναι μια ελπίδα ειρήνευσης στο Αφγανιστάν και μια απόδειξη ότι η συνεχής δέσμευση και προσπάθεια μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα. Εκτιμούμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρήνευση στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ θερμός. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε την εξοχότητά σας για τα σχόλια αυτά. Θέλετε να απαντάτε σε μία-μία ερώτηση ή θέλετε να ακούσουμε περισσότερες. Όπως θέλετε, Πρόεδρε. Ωραία, ας ακούσουμε ένα πρώτο γύρο των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Μίχελ Γκάλα, μέχρι τις 11.30 θυμίζω συνάδελφοι έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Γκάλα, είμαι εδώ στα δεξιά. Σας καλωσορίζουμε κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, εγώ παρακολουθώ τακτικά το Αλτζαζίρα, το αγγλόφωνο Αλτζαζίρα και από το κανάλι αυτό θα μπορούσα να σας πω ότι αισθάνομαι καλά ενημερωμένος. Θα το θέσω έτσι. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την συνεισφορά αυτού του τηλεοπτικού δικτύου και μου αρέσει πάρα πολύ και η αερομεταφορία σας πραγματικά, τέλος πάντων αυτά επί προσωπικού, για τα πολιτικά θέματα. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι εξελίξεις στη σχέση σας με τους Άραβες γειτονές σας και με το Ιράν αν αντιλαμβανόμαστε την σημερινή κατάσταση, την καταλαβαίνουμε. Εσείς βλέπετε κάποιο διέξοδο. Κάποια διέξοδο, με συγχωρείτε. Μπορείτε να φανταστείτε ότι κάποια διαμοσολάβηση εξωτερική θα μπορούσε να είναι επιτυχής. Επίσης, οι σημερινές εμπορικές ροές για σας πώς είναι, είναι όλες μέσω του ενέργειου χώρου του Ιράν. Έχετε δυνατότητα παράκαμψης για τα αγαθά που εισέρχονται σε εσά. Και για τη Λιβύη μια ερώτηση. Εσείς ποιον υποστηρίζετε στην εκεί αντιπαράθεση, γιατί ακούμε νέα διαρκώς ε, για υποστήριξη του Κατάρ προς την τάδε ή τη δύνα πλευρά. Επίσης, γνωρίζουμε ότι έχετε δεσμευθεί με την Ουνρα το οποίο χαιρετίζουμε, Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι θα εξακολουθείτε να την υποστηρίζετε χρηματοδοτικά όπως έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Μαρία Ρένα από πλευράς S&D. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχουμε πολύ στενές σχέσεις στην Υποεπιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και με το Κατάρ έχουμε υπογράψει και μια εταιρική σχέση και σύμβαση με το Κατάρ η οποία μας ικανοποιεί. Μα εξέπλεξε όμω η νέα νομοθεσία σχετικά με την ελευθερία έκφραση στο Κατάρ με υποχώρηση, νέα υποχώρηση, περιορισμό της ελευθερία αυτή. για ανθρώπου ε, που θα είχαν καταδικαστεί ότι έχουν επικρίνει δημόσια τη χώρα τους είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό της χώρας με ποινές φυλάκισης 3 έως 5 έτη θεωρώ ότι αυτό το νέο νομοθέτημα είναι αρνητικό μήνυμα για την ελευθερία έκφρασης ε, στη χώρα σας και θα ήθελα να σας μεταφέρω την ε, έντονη έκπληξή μας και την δυσκολία να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε επικοδομητικά σε πλαίσια θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε την κυρία Αγενά, Ρινιού. Ναταλή Λουαζού. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον ε, κύριο Υπουργό που είναι μαζί μας σήμερα. Είσαι ό,τι αφορά στην ε, διπλωματία του Κατάρι ε, είστε πολύ ενεργητικοί σε διάφορα μέτωπα και σε μια περιοχή κρίσιμη σημασία για εμάς που είναι το Σαχέλ. Στο φόρουμ της Ντόχα, μεταξύ άλλων, αναζητούμε λύσεις μη στρατιωτικής φύσεως ε, για την περιοχή του Σαχέλα και σίγουρα θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για τη σημασία της ε, ε, επανεγκατάστασης του ρόλου των κρατών στην περιοχή αυτή. Έχουμε ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή αυτή. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε μια μάστιγα για την ειρήνευση ε, και της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρη που είναι ο τζιχαντισμός. Οι τρομοκρατικές ομάδες, ποια είναι η ακριβής τοποθέτηση του Κατάρ για τις τζιχαντιστικές ομάδες που διαστριοποιούνται στο Σαχέλ. Μπορείτε να, να καταδικάσετε τις ενέργειές τους όπως το κάνουμε και εμείς. Και αυτές οι υπόνοιες ότι υπάρχει ανεπίσημη χρηματοδότηση από το Κατάρ Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι είναι λανθασμένες και ότι δεν υπάρχει τέτοια χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ κυρία Λουαζό, ID ο κύριος Μαριανή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είμαι εδώ. Ε, έχω, είμαι διστακτικός προς την ε, χώρα σας. Υπάρχει μια ελκυστική πλευρά, σύγχρονη, μεταρρυθμιστική, αλλά αν είναι να πιστέψουμε και κάποιες πηγές ε, πρόσφατες ε, στη Γαλλία, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Δηλαδή ότι έχετε χρηματοδοτήσει τρομοκρατικές ομάδες στη Συρία. Λένε επίσης ότι ήσασταν στο πλευρό των Αμερικανών, ε, των Τούρκων και της Σαουδικής Αραβίας στην όλη αυτή επιχείρηση. Οπότε η πρώτη μου ερώτηση είναι τι πραγματικά έχετε χρηματοδοτήσει εσείς στη Συρία θα συνεχίσετε να το κάνετε. Και σήμερα πώς τοποθετήσετε απέναντι στο ζήτημα της Συρίας. Το δεύτερο, όπως είπε και η κυρία Αινά, υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία έκφραση στη χώρα σας που είναι λυπηρό γιατί έχετε εκδηλώσεις για την ελευθερία του τύπου, τον οποίον τύπο περιορίζεται στη χώρα σας. Επομένως υπάρχει μια ανθιπλή γλώσσα μια διπλή διατύπωση. Θα ήθελα λοιπόν πάρα πολύ να σας ακούσω σχετικά με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δράσεων στη Συρία, όπως και αυτό που ρώτησε η κυρία Λουαζού. Την, τρομοκράτηση, την ε, χρηματοδότηση με συγχωρείτε, τρομοκρατικών ομάδων στη Σαχέλ, όπου έχουμε ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας, κατά κύριο λόγο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαραγιανή. Για τους πρασίνους, η κυρία Λάνζ είπε. Um, θα μιλήσω γερμανικά. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ θα ήθελα να σας απευθύνω το ερώτημα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο τρέχον και ο μελλοντικός σας ρόλος στη Συρία. Δεύτερο ερώτημα. Εσείς μαζί με την, με την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία χαιρετήσατε το ερευνητικό σχέδιο Τραμπ. Γιατί? Ποια είναι τα, τα θετικά στοιχεία? Τι ακριβώς σας έκανε σε αυτό το σχέδιο να το χαιρετήσετε. Ένα ερώτημα λοιπόν για τη Συρία και ένα για το σχέδιο Τραμπ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Κυρία Φωτίγκα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εξοχότατε σας ε, καλωσορίζω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, θέλετε, σας παρακαλώ να μας πείτε την άποψή σας για το σχέδιο Τραμπ για την ε, Μέση Ανατολή για να δοθεί μια διέξοδος στην κατάσταση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις Παλαιστίνης-Ισραήλ. Και επίσης, μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας όσον αφορά τη στάση των άλλων χωρών του κόλπου για το ίδιο αυτό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βιλανοέβα εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Η ποινικοποίηση της διαδήλωσης είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε σε διάφορες χώρες επί τη βάση καταπίεσης και νομοθεσίας. Και εμείς εκφράζουμε λοιπόν την ανησυχία μας για την περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που λαμβάνει χώρα στο Κατάρ. Η απόσυρση της ε, υποστήριξης ε, για τους πρόσφυγες ε, στην Παλαιστίνη αντικαταστάθηκε από το Κατάρ ως παρουσία χρηματοδοτική. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντική συνεισφορά. Από το 49 έχουμε το πρόβλημα της χρηματοδότησης των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στην Παλαιστίνη προσπαθώντας να αποφύγουμε την επιστροφή των ε, προσφύγων. Αυτή, αυτό όλο το προσφυγικό ζήτημα και μετά από την υποβολή του περιβόητου σχεδίου του αιώνα του Τράμπα ε, νομίζετε ότι θα μπορέσει να βοηθήσει, να συνεισφέρει προς την ε, επίλυση του ζητήματος. Αυτός ήταν ο πρώτος γύρος. Θα θέλετε να σχολιάσετε επί των ερωτήσεων που ακούστηκαν. Sorry if I miss... Με συγχωρείτε αν παραλείψω κάποιες ερωτήσεις να με ενημερώσετε αν αφήσω κάτι πίσω. Θα προσπαθήσω να δω τα θέματα ένα-ένα. Ξεκινώντας με το θέμα του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου, το εμπάργκο στο Κατάρ, το αποκλεισμό και αυτό σε σχέση με το Ιράν. Καταρχάς, αυτό ο αποκλεισμός ήταν αναπτρεπτικός για όλη την περιοχή. Το Κατάρ ήταν το θύμα αυτού του αποκλεισμού, αυτού του εμπάργου, εδώ και δύο χρόνια τώρα. Έχουμε εκτιμήσει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τον Εμμυρί του Κουβέιτ στο να διαμεσολαβήσει σε αυτή την κρίση για να επιτευχθεί κάποια επίλυση. Ε, είχαμε κάποιες ελπίδες τον Νοέμβριο όταν ξεκινήσαμε κάποια συνομιλία με τους Σαουδάρβες, αλλά δυστυχώς μετά από δύο μήνες είδαμε αναστολή από πλευράς της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να υποδεικνύεται κάποιος λόγος. Ε, συνεχίζουμε να καλωσορίζουμε τις προσπάθειες μέσω της διαμεσολάβησης του Κουβέιτ ε, να επανέλθουν τα κράτη στη Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων για να πετύχουμε κάποια λύση σε αυτή την κρίση. Το Κατάρ αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα ότι αυτός που χάνει είναι η περιφέρεια και ο λαός της περιφέρειας. Δεν θα υπάρχουν νικητές από αυτή την κρίση. Όλοι θα νικήσουμε εάν κατορθώσουμε να επιλύσουμε την κατάσταση με τρόπο που να μας προστατεύει και να μας προασπίζει από τέτοιες συγκρούσεις στην, στο μέλλον. Το κυριότερο θέμα στον κόλπο ανάμεσα στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ε, ελπίζουμε ότι θα ε, ξεκινήσουν να συνομιλούν ε, λογικά για τα προβλήματα και να σταματήσουν να διαδίδουν προπαγάνδα κατά του Κατάρ. Σχετικά με τις σχέσεις με το Ιράν, που είναι και πάλι μια χώρα γείτονα, ε, που υπάρχουν πολλά θέματα επίσης και με τις ΗΠΑ. Το Κατάρ έχει καλή σχέση γειτονίας με το Ιράν. Το Ιράν άνοιξε τον αεροχώρο, τα λιμάνια του, για τον εφοδιασμό των προϊόντων, για την μετάβαση ε, επιβατών ε, και εκτιμούμε αυτές τις προσπάθειες στήριξης από οποιαδήποτε χώρα, ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες ε, του αποκλεισμού. Τώρα, εμείς θέλουμε να δούμε σταθερότητα στην περιοχή, να μην υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στο Ιράν, διότι και η ΙΠΑ είναι ένας από τους στρατηγικούς μας ε, συμμάχους. Το Κατάρ ε, θα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εγκατάσταση, ε, στρατιωτική εγκατάσταση των ΙΠΑ στην περιοχή και έχουμε σχέσεις γειτονίας και με το Ιράν από την άλλη πλευρά δούλεψαν πολύ σκληρά ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης και της κλιμάκωσής της. Ε, συνομιλήσαμε με όλα τα μέρη, ε, προς τους Αμερικανούς, προς τους Ιρανούς για, και για να προσφύγουν σε διπλωματικές λύσεις και συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι αυτό θα επιληθεί με τη διπλωματική οδό. Υπήρχε και μια ερώτηση για το πώς πάνε τα πράγματα με το εμπόριο τα αεροσκάφη μας ε, πετάνε πάνω τον Ιρανικό χώρο. Υπάρχουν και άλλα που πάνε κατευθείαν από το Κατάρ στο ε, Κουβέιτ ε, πάνω από τον Ιρακινό χώρο. Ο εφαδιασμός γίνεται είτε με αεροπλάνα <clears throat> είτε διαθαλάσσεις που τα λαμβάνουμε στο λιμάνι Χαμίτ το οποίο από το εμπάρκο έχουμε ανοίξει αυτό το λιμάνι και έχει περίπου 27% του εμπορίου της ε, περιοχής και ε, προσβλέπουμε στην επέκτασή του. Βέβαια, αυτή η κρίση θα τερματιστεί, ελπίζουμε, ε, και θα ανοίξουμε διάπλους εμπορίου και θα δούμε την περιοχή να ανθεί περισσότερο σε ό,τι αφορά το εμπόριο μελλοντικά. Σχετικά με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ και το νόμο που, στο οποίο αναφερθήκατε σχετικά με ότι ε, λέτε ότι στοχεύει την ελευθερία της έκφρασης, αυτό δεν ήταν ποτέ πρόθεση του Κατάρ να στοχεύσουμε την ελευθερία της έκφρασης. Είμαστε υπέρμαχοι της προστασία της ε, ελευθερίας έκφρασης στο Κατάρ και ε, συγχωρούμε υπέρ της ελευθερίας έκφρασης για εκτός Κατάρ. Δυστυχώς έγινε κάποια παρερμηνία ότι αυτός ο νόμος ε, στοχεύει την παραπληροφόρηση και όχι την ελευθερία της έκφρασης. Η παραπληροφόρηση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν συμβαίνει μόνο στο Κατάρ και την περιφέρειά μας, συμβαίνει παντού στον κόσμο και ως απόδειξη αυτού ότι αυτό δεν στοχεύει την κριτική. Αυτός ο νόμος επικρίθηκε στο Κατάρ και κανείς δεν έχει ε, προσαχθεί ενώπιν της δικαιοσύνης. Γι' αυτό το, το κάνουμε για να προστατέψουμε τη χώρα μας από την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση που δυστυχώς ξεκίνησε από τότε που επιβλήθηκε ε, το εμπάρκο κατά του Κατάρ. Σας ε, διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση ε, να σταματήσουμε την ελευθερία της έκφρασης και καλωσορίζω οποιαδήποτε σχόλια, αν υπάρχει τρόπος να βελτιώσουμε την κατάσταση και παραμένουμε προσιλωμένοι σε αυτό. Τώρα, σχετικά με τα περιφερειακά θέματα. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω με τη Λιβύη. Το Κατάρ είχε σταθερή θέση από το 2015 ότι η μόνη διάβλη επικοινωνίας και η μόνη στήριξη θα γίνεται μέσω της νόμιμης κυβέρνησης που αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Διεθνή Κοινότητα. Παραμένουμε σταθεροί σε αυτή τη θέση και συνεχίζουμε της ε, συνομιλίας και την επικοινωνία μας ε, ε, με το GNA και καταδικάζουμε κάθε στρατιωτική επιχείρηση από μέρους του στρατηγού Χαφταρ και έχουμε κάνει το γύρο του κόσμου και λέμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και θα πρέπει να υποστηρίξουμε την κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη και να ε, επανέλθει η πολιτική λύση εκεί. Βλέπουμε ότι η διεθνή κοινότητα έχει κινητοποιηθεί εδώ και μήνες, ε, μετά από μήνες ε, μετά από μήνες στην Τρίπολη, αλλά παρακολουθούμε στενά ε, ένα μέρος το οποίο δεν σέβεται τα ψηφίσματα της διεθνούς κοινότητας και παραβιάζει ε, και η κατάπεση του πυρός έχει ε, συμφωνηθεί στη Μόσα, στο Βερολίνο, έχει επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά αυτά δεν έχουν τύχει ε, σεβασμού. Ε, Χθε το λιμάνι της Τρίπολης ε, βομβαρδίστηκε και πριν από μερικές μέρες είχε βομβαρδισμό στο αεροδρόμιο από τον Χαφτάρ και δεν έχουμε δει καμία δράση εναντίον αυτό. Θα πρέπει να σταματήσει το εμπάρκο των όπλων ε, θα πρέπει να σταματήσουν οι ξένες παρεμβάσεις, θα πρέπει να καθίσουν τα μέρη γύρω από το τραπέζι και να συζητήσουν για ε, την, δική τους μοίρα. Ε, είμαστε υποστηριχτές της διαδικασίας και της έκβασης της διαδικασίας του Βερολίνου. Φτάνει να φτάσει σε σταθερότητα στην Λιβύη. Σχετικά τώρα με το Παλαιστινιακό και την στήριξή μας ε, προς την Άνρουα. Το Κατάρ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Παλαιστινιακού λαού και συνείσφερε ε, είτε μέσω από τους οργανισμούς του ΟΗΕ, είτε μέσω από τα προγράμματα που κάνουμε από κοινού με ε, τους του ΟΗΕ. Το Κατάρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές του Άνερουα για να διαφορώσουμε αυτό το κενό που έμεινε μετά από την απόσυρση της αμερικανικής στήριξης στην Άνερουα και πιστεύουμε ότι ο λόγος που η Άνερουα παραμένει ε, ένα σημαντικό φορέα εκεί και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι πρόσφυγε χρειάζονται ε, την βοήθεια του Άνουρα και αυτό είναι σημαντικό. Για... Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το δικαίωμα επιστροφής στη χώρα τους. Έχουμε και σχέδια επίσης ε, να ε, υλοποιήσουμε σχέδια στη Λωρίδα της Γάζας ε, με την ανέγερση κατοικιών, σχολείων για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, ε, παροχή καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα στη λωρίδα της Γάζας. Ε, τώρα εδώ και 18 μήνες αυξήσαμε ε, την παροχή ηλεκτρισμού από δύο ώρες, τώρα είναι γύρω στις 8 ώρες καθημερινά και συνεχίζουμε την παροχή των ε, ηλεκτρικού ρεύματος ε, στη Λωρίδα της Γάζας. Σχετικά τώρα με το σχέδιο Τραμπ ε, στο Μεσανατολικό, εμείς καλωσορίζουμε κάθε πρωτοβουλία που προτείνει, ένα σχέδιο επίλυσης του, της Ισραηλο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης, αυτό πρέπει να συνάδει με την διεθνή νομιμότητα. Και ήταν η θέση του Κατάρ. Εμείς δουλεύουμε με την Αμερικανική κυβέρνηση, ενθαρρύνουμε τους Παλαιστινίου και τους Ισραηλινούς να ε, ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις και θέλουμε ε, στην τελική να υπάρχει ειρήνη ανάμεσά τους αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι οι αραβικές χώρες έχουν συμφωνήσει σε μια πρωτοβουλία αραβικής ειρήνης και έχουν ε, προτείνει αυτή την πρωτοβουλία και αυτό είναι μια δίκαιη βάση επίσης για τις διαπραγματεύσεις. Θα συνεχίσουμε και εμείς να παρέχουμε συμβουλές προς όλα τα μέρη. Θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τους Παλαιστινίους ε, να, ε, και, να ενθαρρύνουμε τις ΗΠΑ να ε, συνεργαστούν με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να δουν ποια είναι τα κενά και τα σχέδια και για ε, να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση. Τώρα, σχετικά με το θέμα της Συρίας, Πιστεύω ότι ένα από τα μέλη σας εδώ τόνισε το ρόλο του Κατάρ στη Συρία ε, που το Κατάρ ε, ε, έχει χρηματοδοτήσει τρομοκρατικές ομάδες στη Συρία. Όχι, η απάντηση είναι ότι ποτέ δεν έχουμε χρηματοδοτήσει τρομοκρατικές ομάδες στη Συρία. Το έχουμε καταστήσει σαφές αυτό. Η στήριξη μας πάει κατευθείαν στο Συριακό λαό, είτε μέσω ανθρωπιστικής στήριξης, είτε μέσω των ανθρωπιστικών οργανισμών, μαζί με τον ΟΗΕ. Τους παρέχουμε αναπτυξιακή βοήθεια, βοήθεια στο τομέα της εκπαίδευσης, πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά ε, στους ε, καταβλισμούς των προσφύγων ε, εποφελούνται της βοήθειάς μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. σε κάποια στιγμή, όταν η στήριξη πήγε προς την αντιπολίτευση, έγινε μια συλλογική προσπάθεια από όλους την ομάδα των φίλων και μαζί με τους άλλους ε, διασφαλίσουμε ότι αυτή η συνεισφορά έγινε ε, ισότιμα σε όλη τη χώρα και προσέχουμε να μην διοχετευτούν χρήματα σε τρομοκρατικές ομάδες και καταγγέλουμε αυτές τις δραστηριότητε. Αυτοί οι τρομοκράτες που βρίσκονται στη Συρία προσπάθησαν να ε, χρησιμοποιήσουν αυτό ως πρόσχημα. Εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες του Συριακού λαού ε, και καταδικάζουμε το, το καθεστώς που δολοφονεί το λαό εδώ και χρόνια και δυστυχώς η διεθνής κοινότητα δεν κατόρθωσε όλα αυτά τα χρόνια να σώσει το σειρακό λαό. Τώρα, σχετικά με το ρόλο του Κατάρ στο Σαχέλ, και ποια είναι η θέση του Κατάρ σε σχέση με του τζιχαζιτζές και πάλι εμείς καταδικάζουμε τις δραστηριότητες τους, τις ενέργειές τους. Θα μπορείτε να δείτε τις θέσεις του κατά, τις έχουμε εκφράσει σαφέστατα. Όλες οι επιχείρησεις που ε, αναλαμβάνονται από τους τζιχαντιστές στο Σαχέλ ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου, τις έχουμε καταδικάσει επίσημα σε δηλώσεις. Εμείς στηρίζουμε τις χώρες του Σαχέλ κατευθείαν και άμεσα με τη στήριξη ε, να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στο Μαλί, στην Πουρκίνα Φασό και άλλες χώρες της περιοχής του Σαχέλ. Το Κατάρ θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις χώρες και να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να ε, επιφέρουν μεταρρυθμίσεις στις δικές τους κυβερνήσεις έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη σταθερότητα στις χώρες αυτές. Νομίζω ότι έχω καλύψει τα περισσότερα ερωτήματα. Συνάδελφοι, έχουμε πέντε λεπτά ακόμα. Εγώ πολύ θα ήθελα να δώσω το λόγο και σε άλλους ομιλητές, αλλά πολύ σύντομα παρακαλώ. Η ε, κυρία Ζόφκο. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ τον Υπουργό. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κατάρ για όλα αυτά που κάνει στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της απορριζοσπαστικοποίησης εννοεί η ομιλήτρια. Είχαμε ένα θέμα με το Αλτζαζίρα <clears throat> που ανέφερε λανθασμένα ε, για κάποια από τα τεκτενόμενα στην Βοσνία Ερζεγοβίνη και γενικώ για την κατάσταση των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, αυτό ε, στο πλαίσιο της ε, καταπολέμησής μας των fake news στα Δυτικά Βαλκάνια, των ξένων μαχητών και κατά κεφαλήν έχετε τους περισσότερους ξένους μαχητές σε αυτή την περιοχή. Μήπως μπορείτε να μας καλύψετε. Η κυρία Καηλή, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ μόλις επέστρεψα από την Ντόχα, όπου είχε ένα, είχατε ένα φόρουμ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για ξένες χώρες που παρεμβαίνουν στην παραπληροφόρηση. Εξεπλάγει από την πρόοδο με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το θέμα των γυναικών που έχετε σημειώσει κάποια πρόοδο. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω με το εμπάργκο ποια είναι ακριβώς η κατάσταση γιατί είχαν υπάρξει συλλήψεις, είχαν υπάρξει και εκτελέσεις δημοσιογράφων σε Σαουδική Αραβία και έχουν ακουστεί διάφορες επικρίσεις και διάφορα σχόλια σχετικά με το εμπάργκο. Μήπως μπορείτε να μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κυρία Ρις. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε τηλεγραφικά καθότι δεν έχουμε χρόνο. Δύο ερωτήσεις κύριε Υπουργέ. Το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου σε δύο χρόνια. Ε, πώς είναι οι συνθήκες ε, εργασίας των μεταναστών εργατών γιατί έχουν γίνει καταγγελίες από πολλές και διάφορες οργανώσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ξέρω ότι οι αρχές του Κατάρ μαζί με τη FIFA είχαν καταλογοποιήσει διάφορα μέτρα τα οποία υποτίθεται ότι υλοποιούνται 22 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιανουάριο αναφέρθηκαν. Πώς πάνε αυτά τα μέσα, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες αυτών των εργαζομένων, που ήταν αρκετά λυπηρές. Επίσης, ε, υπό την έννοια του περιβάλλοντος, γιατί είμαι και από την Επιτροπή για τα θέματα περιβάλλοντος, ε, εσείς αναφέρεστε σε ε, μια οικονομία ουδέτερη στον άνθρακα. Εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς θα μπορούσατε να το πετύχετε. Έχετε προχωρήσει, έχετε ένα σχέδιο πολύ φιλόδοξο για τα φωτοβολταϊκά για δύο χρόνια, αυτά είναι αύριο που λέμε. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο Ο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής είναι εδώ απ' έξω. Αν μπορείτε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, κύριε Υπουργέ, για να πάμε στο επόμενο σημείο, να μην, έχουμε τον, να μην περιμένει ο φιλοξενούμενός μας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, για το Al Jazeera, για τα Δυτικά Βαλκάνια. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε ποιος είναι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Εμείς στο Κατάρ εξασφαλίζουμε να είναι ελεύθερα τα μέσα ενημέρωσης, ανοιχτά για όλους. Όλοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί με το τηλεοπτικό δίκτυο αυτό. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε στην πολιτική του δικτύου. Ε, αν το κάναμε ίσως και να μην είχαμε κάποια από τα προβλήματα που έχουμε με τα κράτη εμπάργκο, αλλά τέλος πάντων το Al Jazeera έχει τη δική τους επαγγελματική ομάδα, μπορεί να λάβει οποιονδήποτε διάλογο. Σας καλώ λοιπόν να έρθετε στο Κατάρ, να δείτε από κοντά ποια είναι η πρόοδος και ίσως να βρείτε και την ευκαιρία να τους μιλήσετε απευθείας. Ε, για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για τις προετοιμασίες του παγκοσμίου κυπέλου, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Ο ILO έχει γραφεία επιτόπου. Έχουμε βελτιώσει και την ικανότητα διαφόρων κρατικών φορέων να υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές νομίζω ότι έχουν αποτυπωθεί στην εξέλιξη των έργων προετοιμασίας και δεν δεχόμαστε καμία κατάχρηση ή παραβίαση των δικαιωμάτων των φιλοξενωμένων εργαζομένων για τις εγκαταστάσεις του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα, για την ε, ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα για το παγκοσμίο κυπέλο. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο για τα θέματα κλιματικής αλλαγής και ουδετερότητας άνθρακα. Οικοδομούμε ένα μία από τις μεγαλύτερες ηλιακές μονάδες παραγωγής ενέργειας. Δεν είμαι βέβαιος για τα ακριβή μεγέθη, αλλά αυτά που είχαμε από τις προηγούμενες εκθέσεις λένε ότι έχουμε ήδη υπερβεί τις δεσμεύσεις, τους στόχους που είχαμε τοποθετήσει. Όλα τα στάδια έχουν οικοδομηθεί ώστε να είναι περιβαλλοντικά φιλικά και να μειώνουν το αποτύπωμα του άνθρακά τους για το καθεστώς του εμπάργου. Μίλησα και νωρίτερα για αυτό. Ε, ελπίζουμε όλοι οι ενεχόμενοι να ξαναδούν τη λογική, να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει μια, ένας συνολικός παρανομαστής που μπορεί να δώσει αριθμητική απάντηση στα πάντα. Ε, υπάρχουν διάφορες συνιστώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ελπίζουμε, ελπίζω αυτή η απάντηση να σας καλύπτει και ελπίζουμε και εμείς να δούμε σύντομα λύσεις στο θέμα αυτό. Εξοχότητα, ευχαριστούμε πολύ λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε για την ανταλλαγή απόψεων, καλή επιστροφή και θα σας δούμε σύντομα στην Επιτροπή μας και πάλι. Thank you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 taking break, huh? <laughs> Colleagues, without... Συνάδελφοι, χωρίς άλλη καθυστέρηση, λέω να συνεχίσουμε. Καθίστε σας παρακαλώ. Για να περάσουμε στη συζήτηση του σημείου 7. Καλωσορίζουμε θερμά τον εξοχότατο Ριάντ Αλμαλίκη, Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστίνης. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Νομίζω η τελευταία φορά που ήσασταν εδώ μαζί μας ήταν το 2016-2017, όταν ο Έλμαρ Μπρόκ ήταν ε, πρόεδρος εδώ της Επιτροπής. Να, ευχαρισ... να ε, καλωσορίσω επίσης τον πρέσβη, τον κύριο Ραχίμ Αλφάρα, τη Παλαιστίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Βρίσκεστε εδώ για διαβουλεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και το μέλλον τη ε, ειρηνευτική διαδικασία τη Μέσα Ανατολή. Ε, Σα έχουμε μαζί μα εδώ για να μα παρουσιάσετε την άποψη τη Παλαιστινιακή Αρχή σχετικά με αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και θα θέλαμε επίση να συζητήσουμε και το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αναζωογόνηση τη ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και την δημιουργία των προποθέσεων για εκ νέου συνομιλίε Ισραήλ-Παλαιστινιακή Αρχή. Είχαμε μόλι μαζί μα τον πρέσβη του Κατάρ, ε, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Κατάρ, συγγνώμη, και θα έχουμε μαζί μας και τον πρέσβη του Ισραήλ ακριβώς μετά από εσάς. Σας δίνω το λόγο για 10 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σας ευχαριστώ που με υποδέχεστε σε αυτό το κρίσιμο σημείο που μπορούμε να προχωρήσουμε αποφασιστικά προς τα εμπρό για να επιτύχουμε την ειρήνη. Να δώσουμε ένα τέρμα στην σύγκρουση και να την αποφύγουμε για τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί πρέπει να σας ενδιαφέρει αυτό. Κάποιοι ε, ενδεχομένως μπορεί να ισχυρίζονται ότι υπάρχουν πιο πιεστικές συγκρούσεις με πιο άμεσες επιπτώσεις στην Ευρώπη. Κάποιοι ενδεχομένως πιστεύουν ότι η Ευρώπη δεν έχει τη δύναμη να ενεργοποιήσει και να προκαλέσει πραγματική αλλαγή. Γιατί λοιπόν να καταβάλλετε την οποιαδήποτε προσπάθεια. Εγώ δηλώνω ότι η μοίρα ενός έθνους που βασανίζεται και υποφέρει από τον εκτοπισμό εδώ και ε, αιώνες, αξίζει της προσοχής σας. Θέλω να σας δείξω πώς βάσει σχεδιασμού η κατοχή του Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε αποσκοπούσε στην εξασφάλιση του περιορισμού των Παλαιστινίων σε περιοχές όπου ήδη ζούσαν και την επέκταση των επίκων του Ισραήλ στα κατεχόμενα με σαφή στόχο να αρπαγεί η γη και να μειωθεί ο αριθμός των Παλαιστινίων. Αυτό έχει όνομα. Απικιοκρατία λέγεται. Ένα από τα πιο αποτρόπαια φαινόμενα της ανθρώπινης ιστορίας. Να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για την πλέον παρατεταμένη ε, κρίση ασφαλείας από την ίδρωση του ΟΗΕ και η πλέον παρατεταμένη κρίση προσφύγων, η μεγαλύτερη σε διάρκεια κατοχή στην σύγχρονη ιστορία. Να σας πω ότι η Ιερουσαλήμ θα έχει πάντοτε ειδική θέση στο μυαλό και στην καρδιά όλων των ανθρώπων, όλων των θρησκειών και ο θρίαμβος της συνύπαρξης εκεί μπορεί να βοηθήσει στη συνύπαρξη οπουδήποτε στον κόσμο. Να σας πω επίσης, αν σας ενδιαφέρει το, το Ισραήλ, πρέπει να το βοηθήσετε να απελευθερώσει τον εαυτό του από την ιδιότητα της δύναμης κατοχής που ασκεί έλεγχο και εξουσία πάνω σε εκατομμύρια ανθρώπους, τους Παλαιστίνιους. Όμως, αν όλα αυτά δεν αρκούν, θα πρέπει να σας ενδιαφέρει ως προς το τι ανέχεστε σήμερα, γιατί αυτά που ανέχεστε σήμερα μπορούν να διαμορφώσουν τον κόσμο του μέλλοντος. Και στο μέλλον θα έχουμε γίνει μάρτυρες της αποδιάρθρωσης του διεθνούς δικαίου και των πολυμερών κανόνων και της διεθνούς τάξης βάση της πολυμέρειας. Κανόνες που έχουν θεσπιστεί ακριβώς για τις δύσκολες εποχές όπως αυτή που διανύουμε σήμερα. Αυτοί οι κανόνες είναι, εξίσου, είναι τόσο ισχυροί όσο εμείς το επιδιώκουμε. Αν εμείς υποχωρήσουμε θα καταρρεύσουν οι κανόνες. Αν όμως εμείς τους υπερασπιστούμε μπορούν οι κανόνες να μας υπερασπιστούν και να μας προστατεύσουν για πολλές ακόμη γενιές. Η ιστορία διδάσκει στην Ευρώπη τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι στις καλύτερες στιγμές τους και στις χειρότερες στιγμές τους. Σας διδάσκει πόσο σημαντική και πολύτιμη είναι η ειρήνη. Ότι δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο για την ελευθερία. Και ότι η ειρήνη επιτυχάνεται με αμοιβαίο σεβασμό και αξιοπρέπεια. Η ε, ένωσή σας δημιουργήθηκε από ελεύθερα και κυρίαρχα κράτη. Ε, η ελευθερία και η κυριαρχία τους πολλές φορές Επιτεύχθη με μεγάλο κόστος και τίμημα. Κάτι που δεν τους εμπόδισε να συνεργαστούν. Αντιθέτως, τους επέτρεψε να συνεργαστούν. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να σας δώσει μια εικόνα για το πώς μπορεί να ε, επιληθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το σχέδιο τον ΗΠΑ βασίζεται στην ιδέα ότι για να υπάρχει ασφάλεια για το Ισραήλ θα πρέπει εμείς να στερηθούμε την κυριαρχία μας. Αυτό δεν θα επιφέρει ειρήνη. Ούτε θα εξασφαλίσει την ασφάλεια στην περιοχή. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως λύση δύο κρατών. Το σχέδιο αυτό μετατρέπει τα παράνομα τελεσμένα σε πραγματικότητα και μας καλεί να τα αποδεχτούμε. Οι παράνομοι επικισμοί, ο παράνομος πόλεμος, οι παράνομες προσαρτήσεις θα γίνουν η μόνιμη πραγματικότητα της ζωής μας. Δεν δίνει τέρμα στην κατοχή, αντίθετα τη διαονίζει. Το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδιαμόρφωσε την, την διεθνή συνένεση με δύο εθνικές κυρίαρχες ταυτότητες με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ στη βάση των συνόρων το 1969 δεν είναι, δεν είναι συνταγή του παρελθόντος. Είναι ο δρόμος για το μέλλον. Αυτό που είναι λάθος δεν είναι το όραμα. Είναι το γεγονός ότι ότι δεν υποστηρίχτηκε το όραμα αυτό με τα αναγκαία μέσα. Η σημερινή Ισραηλινή κυβέρνηση επέρεται ότι η κατοχή δεν της κοστίζει χρήματα. Μάλιστα παρουσιάζουν και τα ωφέλη αυτής, ενώ εμείς υποφέρουμε από τις δραματικές επιπτώσεις. Ισχυρίζονται ότι εκείνοι μπορεί να ζήσουν μια ομαλή ζωή στα περισσότερα μέρη της χώρας τους για τον περισσότερο καιρό του έτους. Μπορούν να έχουν παρά την κατοχή ομαλές σχέσεις με όλο τον κόσμο. Απολαμβάνουν οικονομική ανάπτυξη κτλ. κτλ. Δεν υπάρχει κανένα τίμημα για το γεγονός ότι χτίζουν παράνομους επικισμούς στις δικές μας ε, εκτάσεις. Ούτε για το ότι σκοτώνουν τους ανθρώπους μας, αρπάζουν τη γη μας, κλέβουν τους πόρους μας, υπαγορεύουν το πώς θα ζήσουμε εμείς τη ζωή μας και κανένας δεν τους βάζει να λογοδοτήσουν. Αυτή η ασυλία των Ισραηλινών έχει δραματικά βλάψει και πλήξει τη ζωή εκατομμυρίων Παλαιστινίων εδώ και δεκαετίες. Όμως άλλαξε και το Ισραήλ, υποσκάπτοντας το στρατόπεδο της, ειρήνης και προωθώντας όλους εκείνους που προωθούν παράνομες δράσεις. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι καλοί φίλοι του Ισραήλ. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Στο βαθμό που αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ μπορεί να χτίζει απικίες στις δικές μας περιοχές, στις δικές μας εκτέσεις ή ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το Ισραήλ μπορεί να έχει ασυλία για τους στρατιώτες τους, τους, επίκες, τους επίκους του που διαπράττουν εγκλήματα πολέμου. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζεται τέτοιες δράσεις. Γνωρίζουν οι φίλοι του Ισραήλ πού θα οδηγήσουν όλα αυτά. Δεν είναι ο δρόμος αυτός για να επιτευχθεί η ειρήνη ούτε για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια οποιοδήποτε προωθεί την ασυλία του Ισραήλ βλάπτει την προοπτική της ειρήνης. Δεν μπορεί κανείς να δικαιολογήσει, να αιτιολογήσει ιστορικά, νομικά ή πολιτικά εγκλήματα εις βάρος παιδιών. Δεν μπορεί κανείς να υποστηρίζει ή να υπερασπίζεται εγκλήματα πολέμου. Δεν μπορεί να μην λογοδοτεί το Ισραήλ. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δίκαιο και δεν υπηρετεί την υπόθεση της ειρήνης. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δραματίσει ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριζε πάντοτε τη λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 1969, σε μια εποχή που η Παλαιστίνη, το Ισραήλ και η ΙΠΑ δεν είχαν υιοθετήσει κανείς τους ένα τέτοιο όραμα. Και όταν τελικά αυτό έγινε συνένεση, αυτό συνέβη και χάρη στη στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εταιρικέ σχέσει και με την Παλαιστίνη και με το Ισραήλ. Έχει κανόνε που προωθούν την ειρήνη και πρέπει να του εφαρμόσει. Το Κοινοβούλιο εδώ έχει τα εργαλεία για να ασκήσει πίεση. Έχει αρμοδιότητες και εξουσίες και από αυτή την άποψη επομίζεται και ευθύνε. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία εξαίρεση για το Ισραήλ. Οι παράνομες δράσεις είναι παράνομες ανεξάρτητα από το ποιο τι διαπράττει. Όποιος κι αν προβαίνει σε τέτοιε πράξεις πρέπει να λογοδοτεί. Αν δεν αναλυφθεί η δράση τώρα, πώς θα αποτρέψουμε το Ισραήλ από το να προσαρτήσει παλαιστινιακές εκτάσεις. Κάτι που έχει γίνει κεντρικό θέμα στις Ισραηλινές εκλογές. Το, συνολικό σύστημα του Ισραήλ βασίζεται στην μη προσβασιμότητα σε συγκεκριμένες περιοχές μέσω της βίας. Και οι προσαρτήσεις είναι η έσχατη έκφραση αυτής της πολιτικής. Η Ευρώπη θα κοιτάξει, θα, θα, κοιτάξει ως άπραγος παρατηρητής ενώ όλα αυτά συμβαίνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει, όχι μόνο γιατί υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, που θα καταστρεφόταν από την προσάρτηση, αλλά και λόγω της αντίθεσής της στην παράνομη προσάρτηση, όχι μόνο στην Παλαιστίνη, οπουδήποτε στον κόσμο. Και καθώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του για να στηρίξει την κατοχή και να επιβάλλει την λύση του ενός κράτους των διακρίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να προωθήσει την λύση των δύο κρατών συμπεριλαμβανομένη αναγνώριση τη Παλαιστίνη στα σύνορα του 69. Μια τέτοια αναγνώριση θα αποτελούσε συμβολή στην ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Αναγνωρίζουμε επίση το μερίδιο ευθύνη μα και τι υποχρεώσει που μα ε, επιβαρύνουν όσον αφορά την ε, προώθηση της βίας, της ειρήνης, Εμείς τιμούμε τις δεσμεύσεις που, που έχουμε αναλάβει. Είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων όρων αναφοράς του διεθνούς δικαίου και υπό την αιγίδα της διεθνούς κοινότητας άμεσα. Και όταν λέω άμεσα εννοώ τώρα, άμεσα. Καλούμε από αυτή την άποψη την Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκαλέσει διεθνή σύνοδο κορυφής για να προωθηθεί αυτός ο στόχος. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Μην υποτιμάτε τα όσα μπορείτε να κάνετε εσείς. Μην υποτιμάτε πόσο η δική σας φωνή τελικά έχει σημασία και πόσο εκείνοι που πιστεύουν στην ειρήνη στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ χρειάζεται να την ακούσουν. Πόσο χρειάζονται την υποστήριξή σας. Τώρα περισσότερο από ποτέ. Μην υποτιμάτε τα θύματα που μπορείτε να, αποφύγουμε, να αποφύγετε με την στάση σας και πώς τα πράγματα μπορούν θεμελιωδώς να αλλάξουν τη μοίρα και την κατάσταση της περιοχής μας. Πριν από 75 χρόνια η ανθρωπότητα οικοδόμησε αυτήν την πολυμερή τάξη πραγμάτων για να προωθηθεί η δικαιοσύνη και η ειρήνη. Για να τιμήσει το σύνθημα ποτέ ξανά και για να οικοδομηθεί ένα καλύτερο αύριο η Οικουμενική Χάρτα τον, του ΟΗΕ, οι συμβάσει της, Γενε, της Γενέβης, η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η προοπτική ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου, όλα αυτά πηγάζουν από αυτήν την αρχική ιδέα. Αποτέλεσαν έκφραση του θριάμβου της ανθρωπότητας πάνω στις χειρότερες στιγμές της. Η θυσία αν θυσιαστούν αυτές οι αρχές στην Παλαιστίνη, θα τεθούν σε κίνδυνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Βοηθήστε μας να υποστηρίξουμε, να επιτύχουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, εντός αναγνωρισμένων συνόρων, με αναγνωρισμένα δικαιώματα για τους πολίτες των δύο κρατών. Να είναι οι λαοί ελεύθεροι και όχι ο ένας εις του άλλου ώστε να μπορούν να είναι συνεργάτες, εταίροι, να αλλάξουμε τη, την γειτονιά μας προς το καλύτερο και για πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξοχότατε, Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Έχουμε πολύ για σκέψη και εάν μπορώ να δώσω το λόγο σε όλους τους συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο, αλλά για μέγιστο χρόνο δύο λεπτά ξεκινάμε με ε, τον επικεφαλής ε, της ε, αντιπροσωπείας για, το, για την Παλαιστίνη, τον κύριο Πινέδα. Ξεκινάμε με τις ομάδες. Μιχαήλ Γκάλερ πρώτον. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε, Υπουργέ. Νομίζω οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν ε, λυπηθεί βαθέως ότι αυτή η αμερικανική κυβέρνηση ε, δεν είναι πια ούτε καν έντιμος ε, συνομιλητής, διαμεσολαβητής αυτή την διαμάχη. Φοβάμαι ότι αυτό δεν εξυπηρετεί το μακροχρόνια συμφέροντα ούτε του Ισραήλ ούτε της Παλαιστίνης. Βλέπω προοπτική για δίκαιη λύση μόνο εάν μια μέρα η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί θα συνεργαζόντουσαν με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους προς μια βιώσιμη λύση δύο κρατών. Αυτά που παρουσιάζονται ως σχέδιο από τον πρόεδρο Τραμπ δυστυχώς δεν συμβάλλουν προς κάτι το οποίο ε, μπορεί να αποκαλεστεί ως ένα βήμα προς την ε, ειρήνη. Εάν είμαστε σε αυτή την κατάσταση με την τρέχουσα κυβέρνηση Τραμπ, αναρωτιέμαι ποια είναι η άποψή σας. Πώς θα μπορούσαμε εμείς, τι θα μπορούσαμε εμείς στο μεταξύ ε, τι μέτρα θα μπορούσαμε να λάβουμε για να μετριάσουμε τις δυσκολίες ή να απαλύνουμε την κρίση, τι θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες που εσείς θα προτείνατε στα επόμενα βήματα, εν αναμονή ίσως ε, μιας άλλης πολιτικής από πλευράς Ουάσιγκτον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μιχαήλ Γκάλερ. Μαρία Αρίνα. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την παρέμβασή σας. συμφωνούμε όλοι ότι αυτό το σχέδιο είναι μια πρόκληση προς το Παλαιστινιακό λαό, το έχετε πει εσείς, αλλά θα έλεγα ότι είναι και ύβρις ε, σε διεθνές επίπεδο, ε, προς την πολυμέρεια. Υπάρχουν, σε αυτούς που πιστεύουν στην πραγματική πολυμέρεια και στο διεθνές δίκαιο, στο οποίο ανήκει η Ευρώπη και το οποίο σέβεται. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όμως δεν είναι εδώ. Ε, σήμερα το πρωί είχαμε τον ε, Πρωθυπουργό από το Κατάρ που μας είπε ότι εν τέλει αυτό το σχέδιο θα μπορούσε να συζητηθεί. Εγώ θέτω το ερώτημα, πώς γίνεται η σύμμαχοί σας από τις αραβικές χώρες να ε, μην έχουν μεγαλύτερο λόγο ε, απέναντι σε αυτό το σχέδιο Τραμπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κατάλογος έχει κλείσει των αγοριτών. Προσπαθώ να δώσω το λόγο σε όλους αυτούς που έχουν ε, βάλει έτοιμα ε, να μιλήσουν, αλλά έχουμε κλείσει τον κατάλογο. Ο κύριος Αστέβιτσιος για την ομάδα Renew. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ, ε, αποδεχόμαστε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ε, καθυλωθεί. Δεν επιτελείται καμία πρόοδος ε, μέχρι στιγμής, αλλά πρέπει να είμαστε πιο αισιόδοξοι για τις νέες γενιές, τα παιδιά που μεγαλώνουν σήμερα. Άρα, Υπουργέ, ε, παρακολουθούσα προγράμματα παιδικά στην Παλαιστινιακή τηλεόραση, όπου τους λένε να απαγγέλνουν αντισημιτικά ποίηματα για να δοξάζουν τους μάρτυρες ε, και να καταδικάσουν τους Εβραίους, ε, να τους κατανομάζουν ως τους πιο βάρβαρους λαούς στον κόσμο. Ε, τι είδους γενιά να αναμένουμε να έχουμε στην περιοχή σας, Υπουργέ, όταν αυτά τα παιδιά φτάσουν στην εξουσία και όταν φτάσει η σειρά τους να λάβουν αποφάσεις. Δεν πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα να αναθεωρηθούν ίσως αυτές οι δράσεις προπαγάνδας κατά των Εβραίων για να κτίσετε μια πιο συνεκτική νέα γενιά που να είναι ικανή να απλώσει το χέρι και να καθίσει γύρω από την τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Πέτρας, ε, δεν, έχουμε, δεν έχει ζητηθεί ο λόγος από το ID, η κύριε Λάγκστιν, από τους Πράσινους. <laughs> Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ για τα όσα μας είπατε. Και η δική μου ερώτηση αφορά το σχέδιο Τραμπ, που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ατυχές. Από την άλλη μεριά, αν θέλει κανείς με το ζόρι να το δει θετικά, θα μπορούσε να πει ότι δίνεται μια όθηση στην όλη ε, διαδικασία ειρήνευσης Παλαιστίνης-Ισραήλ, ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις επίκυνται. Ποια είναι η δική σα άποψη. Οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Παλαιστίνης έχουν πλέον αποτύχει θεμελιωδώς. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσουν οι επαφές, οι συνομιλίε. Εγώ θεωρώ ότι σε τελική ανάλυση δεν θα μπορέσει να αποφευχθεί ε, η προοπτική του να δοθεί μια καλή βιώσιμη λύση βάσει των αρχών του διεθνούς δικαίου. Ποια είναι η δική σας άποψη, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επίδραση αυτού του σχεδίου Τραμπ στις μακροπρόθεσμες σχέσεις Παλαιστίνης-Ισραήλ. Ευχαριστώ πολύ για το ECR. Δεν υπάρχει συντονιστής. Δίνω το λόγο στον κύριο Ρόισεν Mr. Ο κύριος Ρόισεν. Είμαι και εδώ ε, επικεφαλής της ε, για την αντιπροσωπεία ε, για το Ισραήλ. Θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους της αντιπροσωπείας. Έχετε το λόγο τώρα. Μιλήστε σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ, είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε μαζί μας, διότι ο διάλογος είναι απαραίτητος. Ο διάλογος μαζί μας είναι απαραίτητος, αλλά και ο διάλογος ανάμεσα στους Παλαιστινίους και το Ισραήλ. Από αυτά που είπατε, κρατώ ότι είστε έτοιμος να διαπραγματευτείτε, το είπατε, ε, εάν το Ισραήλ αποδείξει ότι είναι τέρος για την ειρήνη. Νομίζω είναι κάτι που πάει πιο πέρα από αυτό που ακούσαμε, που ήταν η απόρριψη του σχεδίου ειρήνης που βρισκόταν επιτάπτως προς συζήτηση. Τώρα μιλήσατε για τις βίαιες επιθέσεις στην Γάζα. το Ισραήλ θα πρέπει να προασπιστεί κατά των επιθέσεων στη Γάζα. Είστε διατεθειμένοι και έτοιμοι να αποστασιοποιηθείτε από την, ε, τις βίας πράξεις της Χαμάς από τη Γάζα και είστε διαθετημένος να κάνετε ό,τι μπορείτε να, να διασφαλίσετε ότι οι τρομοκρατικές ομάδες ε, έχουν διαλυθεί. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πορεία της βίας και το τονίζω αυτό ιδιαίτερα διότι χωρίς ε, προϋποθέσεις θα πρέπει να μεταβείτε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Αυτό ε, το έχει πει η διεθνή κοινότητα. Ε, με βάση την έναξη των διαπραγματεύσεων σα δω να μεταβείτε στην τράπεζα και σα ρωτώ αν είστε έτοιμοι να μεταβείτε. Η κυρία Βίλα Νουέβα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, Υπουργέ. είναι μια κατάσταση που δεν πάβει να επιδεινώνεται για, την... για τους Παλαιστινίους με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Το σχέδιο αυτό που... το προσβλητικό αυτό σχέδιο που παρουσιάστηκε επιχειρεί να παρακάμψει απολύτως το διεθνές δίκαιο και έχει και πολύ σημαντικές σοβαρές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον κόσμο ολόκληρο προσπαθεί να νομοποιήσει την προσάρτηση κατεχομένων εδαφών, επικισμών και που ήταν και όλα αυτά το πεδίο το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερη υποστήριξη στην άκρη δεξιά στο Ισραήλ. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα ενιαίο κράτος ανεξάρτητο κάποια στιγμή της Παλαιστίνης χωρίς να έχει συνέχεια εδάφους, συνέχεια υποδομών, οδικών αξώνων κτλ. Πρόκειται για νομιμοποίηση του apartheid που υφίσταται αυτή τη στιγμή και έχει αποκληθεί ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας από το 1973. Ο ύπαντος εκπρόσωπος, ο κύριος Μπορέλ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να θεσπίσει άμεσες σχέσεις με την Παλαιστινιακή πλευρά. Υπό ποιε προποθέσει, κύριε Υπουργέ, νομίζετε ότι θα μπορούσε να λάβει η χώρα ένα τέτοιο διάλογο, μια τέτοια επαφή μαζί με την αρχή σα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Εγώ σας ευχαριστώ για το ΕΛΚΟ, κύριο ο κύριος Μπεσέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, Υπουργέ. Υπουργέ, σας βλέπω σήμερα εξαιρετικά επιθετικό, αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι. Αυτό ακυρώνει οποιαδήποτε προσδοκία ότι θα μπορούσαν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι έχουμε τη μοναδική ελπίδα, ίσως, ε, ίσως μια από τις τελευταίες ελπίδες για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Η Παλαιστίνη θα πρέπει να καταλάβει τις ανάγκες ασφάλειας του Ισραήλ ενό. και βεβαίως το Ισραήλ θα πρέπει να κατανοήσει τις δικές σας ανάγκες. Αλλά το να τηρούμε να τηρείτε η Ισραηλινή θέση όπως τηρείτε παραδιασιακά και τη δική σας θέση ε, χωρίς καμία ευελιξία, δεν θα καταλήξετε σε ειρήνη. δική μου εισήγηση ως πρώην αρχηγός κράτους που αναγνώρισε την Παλαιστίνη ως κράτος, θα πρέπει να διαπραγματευτείτε και να καταλάβετε τα εδαφικά προβλήματα του Ισραήλ που δεν μπορεί να αποδεχτεί αλλαγή της σύνθεσης του πληθυσμού. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσετε. Οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες μπορούν να αλλάξουν τη σύνθεση του πληθυσμού. Εάν θέλετε να συζητήσετε ανοιχτά το θέμα, πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί ε, και η αλλαγή των εδαφών θα πρέπει να συζητηθεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταίοι τρεις ομιλητέ κυρία Ιντσιά. Εγώ σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την παρουσίασή του. Κάτι το οποίο με ενοχλεί ε, άσχημα όταν συζητάμε το θέμα αυτό και τελικά καταλήγουμε στο να είμαστε υπέρ της Παλαιστίνης, υπέρ του Ισραήλ. Δεν μ' αρέσει. Το υπέρ σημαίνει ότι είμαι και εναντίον κάποιου άλλου. Το αν, είμαι υπέρ των Παλαιστινίων σημαίνει είμαι εναντίον του Ισραήλ και αντίθετο, το αντίθετο. αυτό που μου αρέσει συνήθως είναι να είμαστε υπέρ της ειρήνης και όχι αντί της ειρήνης. Και εμείς που πιστεύουμε στην ειρήνη, πιστεύω ότι είναι κόλαφος αυτό το, Τραμπ, το σχέδιο Τραμπ. Γι' αυτό το ερώτημά μου ε, ίσως να απηχώ και ερωτήματα που εκφράστηκαν από προλαλήσαντες συναδέλφους, θα είναι ποιο είναι το επόμενο πρώτο βήμα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο ερώτημα. Ε, δεν σχετίζεται κατευθείαν με το σχέδιο Τραμπ, αλλά σχετίζεται με το θέμα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και αυτό είναι οι εκλογές στην Παλαιστίνη. Πώς ε, φαίνονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή με τις εκλογές. Υπάρχουν οποιοδήποτε φραγμοί, τι εμπόδια υπάρχουν, διότι οι εκλογές είναι σύμβολο της σταθερότητας της δημοκρατίας οποιοδήποτε κράτους ε, στην τελική. Ευχαριστώ, κύριος Βάιμες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών. Στην τελευταία θητεία το Ευρωκοινοβούλιο ε, ενέκρινε ένα ψήφισμα για την ασφαλή ε, επιστροφή των Ισραηλινών πολιτών ε, και την ε, επιστροφή των σωρών των ε, δύο στρατιωτών που κρατούνται από την Χαμάς. Τον Ιούνιο του 2019 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επίση ενέκρινε ένα ψήφασμα 2474 για την προστασία των αμάχων σε ένοπλε ε, συγκρούσει και των αγνοωμένων που επανεπιβιβιώνει την σημασία στο να επιτρέπουμε τις, επιτρόπες, τις, ε, τις να γνωρίζουν για την μοίρα των ε, δικών του. Η Χαμάς κατάφορα παραβιάζει αυτή την κατάσταση. τι κάνει η Παλαιστινική Αρχή για να διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή αυτών των αμάχων που κρατούνται κατά τη θέλησή του στη Γάζα και ε, που ε, στερούνται ε, φροντίδες από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό σε πλήρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και οποιασδήποτε ηθική αξιοπρέπειας. Επίση, τι συμβαίνει για να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των σωρών των Χαντάρ Γκολντέν και Ορών Σόλ που δολοφονήθηκαν και των οποίων οι σωροί έχουν κρατηθεί από την Χαμάς. Ο Μικ Wallace. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, ε, Υπουργέ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι χωρίς τις ευλογίες τον ΗΠΑ. Και πιστεύω ότι οι ΙΠΑ δεν θα μπορούσαν να, δίνουν τέτοια ανεφόρου ε, στήριξη ε, χωρίς την συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά Βλέποντας ε, το πού πρέπει να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς πρέπει να λειτουργήσει προς μια ειρηνευτική λύση, δεν πιστεύετε ότι η λύση δύο κρατών έχει πεθάνει, δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε προς μια λύση ενός κράτους, ισότητα ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, όπου να υπάρχουν ατομικά δικαιώματα για όλους και επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων. Ευχαριστώ. Και για να κλείσουμε, η Ιζαμπέλ Βισελαλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω, αλλά νομίζω έχει τεθεί ερώτηση με εισηγήσεις που θέλω να αφήσω κατά μέρους. Αν μπορείτε να αναπτύξετε τη θέση σας για τη λύση των δύο κρατών. Επίσης, εάν θα μπορούσατε να είσαστε έτοιμοι να δεχτείτε διαπραγματεύσεις άμεσες με το Ισραήλ, χωρίς όρους. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων, μια σωρία ερωτήσεων. Θα σας δώσω το λόγο για 10 έως 15 λεπτά να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο ερώτημα. Ναι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε κατευθείαν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ χωρίς προηγούμενους όρους. Ναι, απόλυτα ναι. Φτάνει βέβαια να ε, στους παλιούς όρους αναφοράς που ήδη έχουν γίνει αποδεκτοί από όλο τον κόσμο. Διεθνές δίκαιο, ψηφίσματα του ΟΗΕ και διεθνή νομιμότητα. Εάν αυτό ισχύει, τότε γιατί όχι. Είμαστε έτοιμοι, αλλά το ερώτημα έχουμε κάποιον εταίρο από πλευρά Ισραήλ. Το αμφιβάλλω. Προσπαθήσαμε εδώ και πολλά χρόνια. Και φαίνεται ότι χάνουμε τις ευκαιρίες. Η λύση δύο έχει πεθάνει φαίνεται ε, ο Νετανιάχου προσπαθεί να σκοτώσει αυτή τη λύση δύο κρατών, δημιουργώντας νέα γεγονότα επί ε, το εδάφους, αλλάζοντας τις καταστάσεις και κάνοντα ό,τι είναι δυνατόν για να σκοτώσει αυτή τη λύση. Ε, φαίνεται ότι μας σωθεί όλους προς μια λύση ενό κράτου. Αλλά αυτή η λύση ενό κράτου είναι καταστρεπτική προ το Ισραήλ καθώς και προς όλους τους άλλους. Γιατί... Γιατί ξέρετε, μήπως ξέρετε, νομίζετε ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει στους Παλαιστινίους σε αυτή τη λύση ενός κράτους να έχουν ίσα δικαιώματα ως ίσοι πολίτες ε, ε, σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Αυτό πρέπει να είναι αστείο. Το Ισραήλ ποτέ δεν θα το επιτρέψει αυτό. Τι θα δούμε λοιπόν ως λύση ενός κράτους. Ένα σύστημα apartheid. Η πραγμάτωση του τι βλέπουμε σήμερα στη Δυτική Όχθη. Ένα σύστημα apartheid. Ένα κράτος με δύο συστήματα. Ένα σύστημα για τους Εβραίου του Ισραήλ και ένα άλλο σύστημα για του Άραβες τη Παλαιστίνης. Αυτό είναι που ισχύει στη Δυτική Όχθη και με το σύστημα του ενό κράτου θα προσπαθήσουν να το νομιμοποιήσουν. Δεν θα το δεχτεί το Ισραήλ, αλλά οθεί προ αυτή τη διακατεύθυνση. Το γεγονό ότι μιλάνε για την προσάρτηση του 33% τη δυτική όχθη, τη Κλαδάς του Ιορδάνη, τη Βόρεια Δυτική Όχθη και του οικισμού, τι κάνουν. Οθούν προ μια λύση ενό κράτου. Αλλά στην τελική τι θα προκύψει θα έχουμε σε αυτή τη λύση ενός κράτους 6,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιους Αράβες και 6,7 εκατομμύρια Ισραηλινούς Εβραίους το πρόβλημα τότε θα είναι δημογραφικής φύσεως. Θα είναι, και θα επανέλθω στο δικό σας ερώτημα, εξοχότατε. Θα είναι δημογραφικής φύσεως και σε χρόνο μηδέν θα είμαστε πλειοψηφία. Σε ένα δημοκρατικό σύστημα ενός κράτους, εμείς θα πρέπει να κυβερνούμε. Και ίσως σε δύο χρόνια ο Πρωθυπουργό αυτού του το λεγόμενου συστήματος ενός κράτους, που θα ονομάζεται Ισραήλ ό,τι θέλετε, θα λέγεται Μουχάμετ. Ε, νομίζετε ότι θα αποδεχτεί το Ισραήλ αυτό το πράγμα. Απόλυτα όχι. Καλύτερα για αυτούς να προσπαθήσουν να διατηρήσουν, να προασπίσουν τη λύση δύο κρατών και όχι τη λύση ενός κράτους. Εάν έχουν κοινή λογική, εάν σκέφτονται ε, επακριβώς, ε, αν έχουν την ειρήνη στο μυαλό τους. The two solution. Η λύση δύο κρατών φυσικά εξακολουθεί να ισχύει. Υπάρχει παγκόσμια συνένεση υπέρ της λύσης δύο κρατών. Θα χάσουμε αυτή την παγκόσμια συνένεση για κάτι το οποίο δεν έχουμε. Εάν αν έχουμε στα χέρια μας αυτή τη λύση δύο κρατών, ας την διατηρήσουμε, ας δουλέψουμε για αυτήν παρά κάτι άλλο το οποίο δεν υπάρχει όλος ο κόσμος σήμερα είναι υπέρ της λύσης δύο κρατών Έχουμε δουλέψει 50 χρόνια για να κτίσουμε αυτή τη συνένεση υπέρ της λύσης δύο κρατών. Μόνο η ΙΠΑ και το Ισραήλ είναι οι μόνες δύο χώρες επί του πλανήτη που είναι εναντίον της λύσης δύο κρατών. Εμείς θα τους επιτρέψουμε να μας νικήσουν, να καταστρέψουν αυτή τη λύση δύο κρατών που, για την οποία υπάρχει διεθνή συνένεση, για κάτι που δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει, προς ένα σύστημα apartheid. Είναι αυτό που θέλουμε. Και είναι γι' αυτό που για να απαντήσω σε πολλές από τις ερωτήσεις. Τι πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να προστατέψουμε αυτή τη λύση δύο κρατών. Θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να διατηρήσουμε αυτή τη λύση δύο κρατών. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να επιβάλλουμε τη λύση δύο κρατών αλλά τι είδους λύση δύο κρατών, όχι αυτή σύμφωνα με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, μια πλήρως κατακαιρματισμένη, αποστρατικοποιημένη, χωρίς ε, κυριαρχία, αλλά μια κυρίαρχη δημοκρατική, ε, ε, ένα κυρίαρχο δημοκρατικό συνεχές κράτος του, της Παλαιστίνης. Αυτό ζητάμε στην λύση των δύο κρατών, όχι οποιοδήποτε άλλο ορισμό της λύσης. Εάν ισχύει αυτό, τότε θα δουλέψουμε γι' αυτό. Έχετε τη δύναμη να το κάνετε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση και εσείς θα δείτε ότι θα έχετε έναν εταίρο με την Παλαιστίνη προς την κατεύθυνση της λύσης δύο κρατών, διότι αυτό είναι το καλύτερο για όλους. Επίσης, εάν μιλάμε για λύση δύο κρατών, και επειδή εσείς ως Ευρωπαίοι έχετε αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ, τι λείπει σε αυτή τον τύπο, σε αυτή τη φόρμουλα. Είναι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, η Ρουμανία αναγνώριση. Υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν αναγνώρισαν ακόμη το κράτος της Παλαιστίνης. Και αν θέλετε να διατηρήσετε τη λύση δύο κρατών, αν θέλετε πράγματι να σταθείτε σταθερά κατά της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, θα πρέπει να μιλήσετε ανοιχτά και να παροτρύνετε τις χώρες σας να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης. Είναι ο μόνος όρος έτσι ώστε να μπορούμε να καθίσουμε επίσης όρις με το κράτος του Ισραήλ στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Αλλιώς μπορείτε να φανταστείτε ε, μας ε, ένα κράτος, ένα, έναν λαό υποκατοχής. Για να φύγω από τη Ραμάλα χρειάζομαι άδεια από τους Ισραηλινούς. Για να πάω στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, να φύγω από τη Ραμάλα χρειάζομαι άδεια από το Ισραήλ. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσεις επί ίσης Θα πρέπει να καθόμαστε επί ίσης ε, με ανεξάρτητα κυρίαρχα κράτη και τότε θα διαπραγματευτούμε επί όλων αυτών των όρων. Αυτό είναι σημαντικό. αλλιώ. ξέρετε, ποια είναι η έκβαση, ποια είναι το αποτέλεσμα. Ξεκινήσαμε από τη Μαδρίτη, ε, τη διάσκεψη της Μαδρίτης, προχωρήσαμε και κοιτάξτε που έχουμε φτάσει τώρα. Πουθενά. Πουθενά. Δεν υπάρχει ισότητα δεν υπάρχει ισοτιμία. Οι Ισραηλινοί είναι η δύναμη κατοχή, έχουν το πάνω χέρι, αποφασίζουν τα πάντα επί τόπου και εμεί οι Παλαιστίνοι υποκατοχή θα πάμε εκεί ε, χωρίς δύναμη. Δεν είναι εφικτό. Δεν είναι ευκαιρία που βασίζεται επίση όρους, επίσης όρους. Εάν θέλουμε να δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι όροι και συνθήκες για τις διαπραγματεύσεις, πρώτον και κύριο είναι οι χώρες που δεν αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης να το πράξουν και να δώσουν όφηση προς αυτό και να καθορίσουν ότι η λύση δύο κρατών είναι καλύτερη φόρμουλα για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Αν καλύτερη για διαπραγματεύσεις θα δείτε ότι οι Παλαιστίνοι αμέσως θα αποδεχτούν την πρόσκλησή σας και θα είναι διατεθειμένοι να καθίσουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων για να διαπραγματευτούν το θέμα αυτό. Ναι, μας ανησυχεί η νέα γενιά και στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Και δουλεύουμε για να καλλιεργήσουμε την ειρήνη στη νέα ε, γενιά. Η ειρήνη που θέλουμε να κτίσουμε είναι για αυτούς. Είναι περισσότερο για αυτούς παρά για μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να δουλέψουμε ε, προς ε, μια δίκαιη ειρήνη. Δίκαιη ειρήνη τι σημαίνει. Σημαίνει τερματισμό της κατοχής. Θα πρέπει οι Παλαιστίνοι να έχουν δικαίωμα στην αυτοκυριαρχία και την ανεξαρτησία. Το Ισραήλ δεν μπορεί να είναι η δύναμη κατοχής και ταυτόχρονα να διακηρύττει ότι είναι δημοκρατική χώρα. Δεν μπορεί να είσαι δημοκρατική χώρα ενώ κατέχεις τα εδάφη και τη ζωή ενός άλλου ε, πληθυσμού και το μέλλον του και την πίστη του. Και εμείς όταν απευθυνόμαστε στις γενιές μας, όταν πάνε στα σχολεία, βλέπουν τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Όταν μετακινούνται από τη μια πλευρά στην άλλη, βλέπουν τους επίκους και τους οικισμούς του Ισραήλ. Όταν ε, στις μετακινήσεις τους βλέπουν το τείχος Αυτές είναι πραγματικότητες που οι νέες γενιές των Παλαιστινίων αντιμετωπίζουν καθημερινά στη ζωή τους. Πώς μπορούσαμε εμείς να τους πείσουμε ότι υπάρχει ευκαιρία για το μέλλον αν δεν διαλύσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που μας χωρίζουν από αυτούς, από τους Ισραηλινούς και να μπορέσουμε να κτίσουμε την ειρήνη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτό είναι πρωτής σημασίας. αλλα τρια τρία-τέσσερα λεπτά. Λέει ο Πρόεδρος, στην τελική ανάλυση δεν λέμε α, όχι απλά για να πούμε όχι. Είμαστε διατεθειμένοι να συμμετέχουμε κάθε φορά που προβάλλεται μια ευκαιρία. Και όταν εμφανίστηκε αυτό το σχέδιο Τραμπ και προσπάθησε να αρνηθεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των Παλαιστινίων ε, στην ιδιότητα του κράτους τους και καταστρέφει το εθνικό αφήγημά τους και τους αφαιρεί το δικαίωμα στο να έχουν το δικό τους κράτος, ένα κυρίαρχο κράτος και δίνει στο Ισραήλ πλήρη έλεγχο ε, στην κυριαρχία τους, στην ασφάλειά τους, την εδαφική τους κυριαρχία και στη γη και στη θάλασσα και στον αέρα. Τι είδους οντότητα θα αποδεχτούν οι Παλαιστίνοι. Πριν από μερικές μέρες ο Νετανιάχου έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα Χαγιούμ του Ισραήλ και κατέστησε πολύ σαφές ότι, ξέρετε, οι όροι που τέθηκαν προς τους Παλαιστινίους θα είναι θαύμα αν θα μπορέσουν να εκπληρώσουν οι Παλαιστίνοι αυτούς τους όρους. Και ακόμη και αν γίνει αυτό το θαύμα και οι Παλαιστίνοι κατορθώσουν να εκπληρώσουν αυτούς τους όρους, τότε οι Ισραηλινοί θα είναι αυτοί που θα καθορίζουν κατά πόσον οι Παλαιστίνοι έχουν δικαίωμα να έχουν τη δική του οντότητα, όχι κράτος ή όχι. Ανά πάσα στιγμή στο μέλλον, ακόμη και αν οι Ισραηλινοί δώσουν το δικαίωμα στους Παλαιστινίου να έχουν αυτή τη δική του οντότητα, μπορούν ανά πάσα στιγμή να ε, εισέλθουν, να εισβάλλουν, να ε, αρπάξουν τα εδάφη του, αν πιστεύουν ότι διακυβεύεται και κινδυνεύει η ασφάλειά του. Ελάτε τώρα ποιος από εσά είναι έτοιμος να είναι πολίτης σε μια τέτοια οντότητα. Κανείς. Σας διαβεβαιώ κανείς. Και κανείς από πλευράς Παλαιστίνης δεν είναι έτοιμος να αποδεχτεί αυτό τον εξευτελισμό. Δεν είμαστε κατώτερα όντα σε σύγκριση με όλους εσάς. Θέλουμε να ε, μας χειρίζονται ως ίσους ανθρώπους, να έχουμε δικαιώματα, αξιοπρέπεια, ελευθερία. Θέλουμε να έχουμε ένα ανεξάρτητο κράτος και έχουμε δεσμευτεί προς ειρήνη με το Ισραήλ. Επί ίσης ώρες. Για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό σας παρακαλώ μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Προσπαθήστε να δράσετε τώρα, προτού είναι πολύ αργά, διότι αν το Ισραήλ υλοποιήσει αυτό το σχέδιο Τραμπ και προβεί στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, τότε εσείς καλωσορίζετε τη βία όχι μόνο στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, αλλά σε ολόκληρη την περιφέρεια. Κάτι το οποίο κανείς δεν θα ήθελε να δει και σίγουρα θέλει να αποτρέψει από το να συμβεί. Σας ευχαριστώ. Ε, εξοχότατε εκ μέρου όλων των συναδέλφων σας ευχαριστούμε για την σημερινή παρουσία σας, για τη σημερινή συζήτηση. Θα διατηρούμε τακτικές επαφές με την αντιπροσωπεία σας. Ε, γνωρίζουμε πόσο κρίσιμη είναι η φάση. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις με μεγάλο ενδιαφέρον. Colleagues. Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας, το τελευταίο σημείο πριν διακόψουμε για το γεύμα, στη μία, λέει ο Πρόεδρος, είναι το υπαριθμόν 8 και καλωσορίζω θερμά τον ε, πρέσβη του Ισραήλ στη Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, τον Αρών Λέσνο Ιλάρ, γνωστό σε πολλούς από εμά. Είχαμε ήδη προσκεκλημένους τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ και στην ίδια καρέκλα που κάθεστε τον Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής. Θέλουμε να ακούσουμε και από εσά βεβαίως την οπτική γωνία του Ισραήλ για την όλη ειρηνευτική διαδικασία και βεβαίως τις ε, πρόσφατες ε, προτάσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ε, θα σας δώσω το λόγο, ήδη πολλοί άριθμοι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή και έχετε το λόγο κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους λέει ο ομιλητής. Έχω μια σύντομη δήλωση. Να σας πω πρώτα απ' όλα όμως κύριε Πρόεδρε ότι σήμερα το πρωί εκπλήρωσα τα, το πολιτιακό μου καθήκον και ψήφισα διότι όλοι οι διπλωματικοί υπάλληλοι ψηφίζουν διαλογραφίας για τις εκλογές που θα λάβουν χώρα σε δύο εβδομάδε και το είπα γιατί βεβαίω είμαι υπερήφανο που συμμετείχα αλλά και επίση επειδή διερχόμαστε μιας ευαίσθητη πολιτικής στιγμής και πρέπει να την προσέξουμε. Να πω καταρχάς κάποια πράγματα για τις σχέσεις Ισραήλ-Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σταθερές, με δυνατότητες, με κοινέ αρχές, κοινέ αξίες και κοινή παράδοση και ιστορία. Θα αναφερθώ απλώς σε δύο περιοχές συνεργασίας μεταξύ του Ισραήλ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα ασφάλειας και ειρήνης και στα θέματα τεχνολογίας και έρευνας, που δείχνουν τα δύο αυτά παραδείγματα. Θα πω απλώς ότι το Δεκέμβριο πέρυσι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας και Κοινοτομίας, με ε, άνοιξε μία έδρα και στο Τελαβίβ. Οι άλλες δύο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στη Silicon Valley και στην Κίνα. Εξωτερικές δηλαδή έδρες. Το οποίο προφανώς μαρτυρεί τις ε, συνεισφορές του Ισραήλ σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το τομέα και την αναγνώρισή του από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωση. Να αναφερθώ στα θέματα ασφαλείας και ειρήνης. Είμαι σίγουρος και ελπίζω ότι μπορούμε μαζί να δουλέψουμε για τα θέματα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή μας και είναι κρίσιμη σημασία η αναγνώριση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης των πολυάριθμων προκλήσεων που έχουμε για την ασφάλεια μας και την ειρήνη στην περιοχή, υπαριθμόν ένα είναι το Ιράν. Γνωρίζω ότι με έχετε προσκαλέσει σήμερα για να μιλήσω για το Παλαιστινιακό, αλλά ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι το Ιράν. Και δεν είναι κίνδυνος μόνο για το Ισραήλ. Το Ιράν απειλεί όλες τις φιλοδυτικές χώρες όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Όπως λοιπόν περιμένετε από εμάς τους Ισραηλινούς να αναγνωρίζουμε και να λαμβάνουμε υπόψη μας τις ευρωπαϊκές ευαισθησίες λέει ο και εμείς το ίδιο περιμένουμε από εσάς. Και όταν μιλάτε για ιρανική απειλή προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια, πρέπει να αντιληφθείτε ότι το Ιράν απειλεί την ίδια την ύπαρξη, λέει ο μιλητής, του κράτους του Ισραήλ και άμεσα και μέσω χρησιμοποίησης αντιπροσώπων. Πρόξεις, για να το πούμε ελληνικά. Τώρα, αυτό που μας οδηγεί στις προσπάθειές μας είναι η ειρήνη με τους γείτονές μας, όλους τους γείτονές μας και τους Παλαιστινίους. Εξασφαλίζοντας βέβαια την ασφάλεια του Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ο μόνος που μπορεί να ορίσει τι είναι προς το συμφέρον της ασφάλειάς του, λέει ο Μιλτής, για την πρόταση του Αμερικανού Πρόεδρου η συμβουλή μου προς όλους εκείνους που ελπίζουν για ειρήνευση στο ζήτημα Ισραήλ-Παλαιστίνης, φαντάζομαι όλους σας εδώ, είναι να εστιαστείτε σε αυτά που κατά την άποψή σας είναι τα θετικά στοιχεία, οι θετικές πτυχές του σχεδίου και θα ενθάρρυνα και τους Παλαιστινίους να κάνουν το ίδιο. Κατά την άποψή μου το σχέδιο έχει μια τέλεια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων του Ισραήλ για ασφάλεια και των προσδοκιών των Παλαιστινίων για ανεξαρτησία. Είναι ένα καλό σχέδιο για την ειρήνη. Ελπίζουμε ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή και θα επαναφέρει τους Παλαιστινίους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τα τελευταία 20 χρόνια, να θυμίσω, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, το Ισραήλ και οι Ηνωμένε Πολιτείε υπέβαλαν προτάσεις στους Παλαιστινίους για ειρηνευτικά σχέδια. Το πιο πρόσφατο ήταν του πρόεδρου Ομπάμα το 2014. Όλα αυτά τα απέρριψαν οι Παλαιστίνοι. Το σχέδιο Τραμπ πηγαίνει στη ρίζα, στο βαθύτερο αιτίο της, της αντιπαράθεσης ότι πρέπει να αναγνωριστεί το Ισραήλ ως το κράτος των Εβραίων. Υπάρχουν εδάφη στην Ιουδαία και στην ε, Σαμάρια που είναι πολύτιμα για την παραδοσή μας, θεμελιώδη και εξετάζει και το καθεστώς εδαφών που δεν θα είναι μέρος τη κρατικής επικράτειας, της εδαφικής με επικράτειας του Ισραήλ στο μέλλον. Προκειμένου να έχουμε ένα μέλλον αξιοπρέπειας, ευημερία και ελπίδα για όλους. Το σχέδιο δίνει αυτή την προοπτική στους Παλαιστινίους. Το σχέδιο δεν εκριζώνει κανέναν, δεν διώχνει κανέναν από τα σπίτια τους. Ούτε Ισραηλινό, ούτε Παλαιστίνιο προτείνει καινοτόμε λύσει, όπου θα έχουμε όμορες περιοχές για να επιτρέπουν ελεύθερη μετακίνηση και συνοδεύεται και από ένα σχέδιο επενδύσεων 50 δισεκατομμυρίων που θα εξασφαλίσει ένα μέλλον ευημερίας για τους Παλαιστινίους. Οι μαζικές αυτές επενδύσεις θα δημιουργούσαν θετική αλλαγή που θα την αισθανόταν θα την έβλεπε κάθε Παλαιστινίος. Τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της χώρας μου, με την διατήρηση του ελέγχου ασφαλείας στο σύνολο της περιοχής δυτικά του Ιορδάνη, δίνοντας μόνιμο ανατολικό σύνορο στο Ισραήλ, για να προστατεύσει το μακρύτερο χερσαίο σύνορό της, είναι κλειδί για την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ. Το σχέδιο επίσης προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατικοποίηση της Γάζας. Αυτό είναι θεμελιώδης σημασίας όχι μόνο για τους Ισραηλινούς αλλά και για τους Παλαιστινίους. Καθιστά σαφές ότι το προσφυγικό πρόβλημα των Παλαιστινίων θα πρέπει να επιληθεί εκτός της εδαφικής επικράτειας του Ισραήλ. Και προβλέπει και την ενωμένη Ιερουσαλήμ υπό Ισραηλινή κυριαρχία με τα κέντρα λατρείας προσβάσιμα για όλους και τη διατήρηση του καθεστώτος του όρους του ναού. Ε, ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι δεν θα χάσουν αυτή την ευκαιρία οι Παλαιστινοί, γιατί είναι ευκαιρία και για τις δύο πλευρές. Το Ισραήλ δεν θα τη χάσει αυτή την ευκαιρία. Και ελπίζουμε να μην τη χάσει αυτή την ευκαιρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μια πραγματική προσδοκία και ελπίδα για όλη την περιοχή. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη για την παρουσίαση των Ισραηλινών απόψεων, ιδίως για τις τελευταίες σας παρατηρήσεις, γιατί αυτά συζητούμε εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όλο το πρωί. Έχω 15 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα προσπαθήσουμε να τον δώσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Βυσλαλίμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Είπατε ότι είστε υπερήφανος που ψηφίσατε σήμερα το πρωί. Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που ζουν σε μια δημοκρατία την ίδια στάση θα έπρεπε να τηρούν και αυτό δεν είναι καθόλου προφανές ε, στον πλανήτη μας σήμερα. Μιλήσατε πολύ για την ειρήνη. Και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι όλοι θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα στην ειρήνη. Και είναι μια μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή που ζείτε. Σας άκουσα να λέτε επίσης ότι η πολιτική του Ιράν είναι μεγάλο πρόβλημα για το Ισραήλ και ότι είναι και για εμάς πρόβλημα. Φαντάζομαι να αντιλαμβάνεστε ότι για εμάς το σχέδιο που προτάθηκε από την Αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να μας βρει απολύτα σύμφωνους. Ενέχει τεράστια προβλήματα για εμάς και θα θέλαμε να μπορούμε να δουλέψουμε επί διαφορετικής βάσης διαπραγμάτευσης. Και θα ήθελα να υποβάλω και σε εσά την ίδια ερώτηση που είχα υποβάλει στον προηγούμενο ομιλητή προσκεκλημένο. Η λύση των δύο κρατών, διότι έχουμε, ε, ε, έχει ακουστεί και το ένα κράτος και τα δύο. Ε, νομίζω ότι είναι κρίσιμο το θέμα, γιατί φοβούμε ότι δεν εννοούμε πάντα το ίδιο πράγμα όταν η μεν ή δεν αναφέρονται στα δύο κράτη. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και εσάς. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Αγενά για το SND. Ε, πάντα διακινδυνεύω να με επικρίνουν αν δεν δώσω, το λόγο στους συντονιστές για το S&D. Κυρία Ρενά, καλώς δεν είναι. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Άκουσα την εισήγηση του κύριε Πρέσβη για το περιεχόμενο του σχεδίου και η ερώτηση μου είναι απλή. Αν αυτό το σχέδιο πράγματι σέβεται και τις δύο οντότητες, γιατί το Συμβουλίο Ασφαλείας ε, δεν το... Μάλλον, γιατί ο κύριος Τραμπ δεν το υπερασπίστηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Γνωρίζετε τις σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ισραήλ επί τη βάση Τη διεθνού συνένεση και επί τη βάση του Διεθνούς Δικαίου και μια σειρά συμβάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει αυτές τις συμβάσεις, επομένως δεσμεύεται νομικά από τις συμβάσεις αυτές. και όταν συνεργαζόμαστε με έναν εταίρο που προφανώ δεν δεσμεύεται τι ε, συμβάσει του διεθνού δικαίου, διότι το σχέδιο Τραμπ δεν συμμορφώνεται προς τις συμβάσεις αυτές. Το κράτος του Ισραήλ είναι έτοιμο να εγκαταλείψει τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα τη συμφωνία σύνδεσης που έχουμε σήμερα ενισχύει. Είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο που διέκοψαν τη σχέση τους μαζί μας ε, και ανέλαβαν τις συνέπειες. Το Ισραήλ, αν σήμερα πει η διεθνή συνένεση δεν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει το σχέδιο Τραμπ, είναι σαν να λέτε δεν μας ενδιαφέρει η συμφωνία σύνδεσης και επομένω αναλαμβάνουμε το τίμημα. Είσαστε έτοιμοι να αναλάβετε αυτό το τίμημα. Σας ρωτώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για το Renew ο κύριος Μπάουσα. Μπάουσα. Μπάουσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ισπανικά, Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον ε, κύριο Πρέσβη που βρίσκεται στην αίθουσα αυτή, στο Κοινοβούλιο, απαντώντας όχι μόνο στα ερωτήματά μας, αλλά αντιμετωπίζοντας και τον καθόλου κρυμμένο αντισημιτισμό που εκφράζουν διάφοροι συνάδελφοι, λέει ο μιλητής. Ήθελα να πω, όπως θα ξέρετε, την περασμένη εβδομάδα η Κλάρα Πονσαντή, που διαφεύγει της Ισπανικής δικαιοσύνης έκανε κάποιες δηλώσεις που δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω, αλλά αναφέρομαι στο περιεχόμενό τους. Και έκανε μια σύγκριση του Ισπανικού κράτους με τον Αδόλφο Χίτλερ. Συνέκρινε μια δικαστική διαδικασία στο ανώτο δικαστήριο στην Ισπανία με το ολοκαύτωμα. Ήθελα να ξέρω τι, πώς σας φαίνεται εσάς μια τέτοια δήλωση, λέει ο μιλητής. Άκουσα τη δήλωσή σας και άκουσα και άλλους ομιλητές να μιλούν για ένα θεμελιώδους σημασίας θέμα ότι το κράτος του Ισραήλ απειλείται με καταστροφή, με αφανισμό από διάφορες εξωτερικές απειλές. Εμείς κύριε Πρέσβη ως Ευρωπαίοι τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να πείσουμε το Ισραήλ ότι ακούμε τις ανησυχίες για την ασφάλεια που έχετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπονφρίσκο εκ μέρους του ID. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, σας άκουσα με, μεγάλη, με μεγάλο ενδιαφέρον. Ασκήσετε και, τα, και το εκλογικό σας δικαίωμα και είστε υπερήφανος. Αυτό είναι κάτι που έχουμε κοινό. Την αγάπη μας για τη δημοκρατία. Εγώ ήδη σε, στην, στις αίθουσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχω ήδη εκφράσει την εκτίμησή μου για το σχέδιο του Τραμπ που επανέφερε στην επικαιρότητα το θέμα της ειρήνευσης του Ισραήλ με την Παλαιστίνη και της ευρύτερης περιοχής. Εγώ θεωρώ ότι η υπεράσπιση της ειρήνης και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από την εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας του Ισραήλ, γιατί σημαίνουν το ίδιο. Και σας ρωτώ με αυτά. Εσείς πιστεύετε ότι το σχέδιο Τραμπ και η δική σας δυνατότητα να ολοκληρώσετε μια ευνοϊκή διαπραγμάτευση για την ειρήνη στην περιοχή θα βοηθούσε και άλλες περιοχές στη Μέση Ανατολή, στην Μεσόγειο, στις γειτονικέ ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνουν ασφαλέστερες για όλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου των Πρασίνων η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια για τη συνάδελφα από το Ρινιού. Ένας φίλος μου από το Ισραήλ στο Ισραήλ μου είπε ότι η κατοχή δεν είναι κόσερ. Ε, αυτή πρέπει να είναι και η αρχή που θα διέπει τη δική μας τάση με βάση το διεθνές δίκαιο. Και να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη απαντήσει. Ο κύριος Μπορέλ σαφέστατα την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο δήλωσε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υποστήριξη των περισσότερων ε, πολιτικών ομάδων γιατί εμείς δεσμευόμαστε σε αυτή την Ένωση από το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσαρμόζουμε ή να το εφαρμόζουμε κάποιες φορές όποτε μας συμφέρει. Όχι, κατοχυρώνεται στη συνθήκη μας. Στο άρθρο 21 της συνθήκης μας θα ε, αναφέρει ότι το διεθνέ δίκαιο και οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας αποτελούν τη βάση για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι φυσικά και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ένα σχέδιο το οποίο στην πραγματικότητα ε, ε, διατηρεί υποστρατιωτικό έλεγχο τους ε, Παλαιστινίου που απελάβνει, προβλέπει την απέλαση μάλλον εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από την, από την Παλαιστίνη και θα βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του Ισραήλ. Φυσικά και είναι όχι από εμά. Βεβαίως κατανοώ ότι θέλετε ειρήνη με τους γειτονέ σα. Όλου μας, μας κινητοποιεί μια τέτοια επιθυμία. Γι' αυτό και θα επαναλάβω αυτό που υπόθηκε το 2003. Το, το σχέδιο του 2003 για την ειρήνευση με την Ανατολική Ιερουσαλήμ στην Παλαιστίνη, σύνορα του 1969, δύο κράτη. Όλα αυτά βρίσκονταν και στην πρόταση της Γενέβης που είχε συζητηθεί λίγα χρόνια νωρίτερα ως βάση των διαπραγματεύσεων και ταυτόχρονα είπαν ότι αν το Ισραήλ δεχτεί αυτό, όλα τα, όλες οι αραβικές χώρες θα το αναγνωρίσουν τελικά. Μέχρι στιγμής μόλις λίγες αραβικές χώρες έχουν ε, αναγνωρίσει το Ισραήλ. Και με, με, με εκπλήσει το γεγονός ότι το Ισραήλ αγνόησε μια τέτοια ευκαιρία. Το ερώτημα το δικό μου σε εσά είναι γιατί αγνοήσατε μια τέτοια προοπτική για την ειρήνευση, για τη χώρα σα και για την Παλαιστίνη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Από το ECR έχω τρει ομιλητέ. Μπορείτε να αποφασίσετε μεταξύ σα ποιο ε, θα τοποθετηθεί εκ μέρου τη ομάδα των ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Είχαμε και κάποιε διαμάχε εδώ με το ECR το πρωί. Α μην επαναληφθούν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, όπως θα κατανοήσατε από τα σχολεία δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τεράστια υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σχέδιο Τραμπ. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι του Τραμπ. Και έπειτα γιατί είναι γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι βάση διαπραγμάτευσης για ένα ειρηνευτικό σχέδιο ειρηνευτικό και για το Ισραήλ. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στον Μπορέλ, ο οποίος μίλησε για το Ιράν. Είδαμε να δολοφονεί το καθεστώς του Ιράν 1500 και άνω πολίτες του, δεν υπήρξε καταδίκη. Συνεχίσαμε να μιλάμε ε, με μια χώρα η οποία επιθυμεί την καταστροφή του Ισραήλ σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Στην Ισπανία έχουμε και μια σοσιαλοκομμουνιστική κυβέρνηση η οποία καθόλου δεν είναι υπέρ του Ισραήλ και έχουμε και δημοτικά συμβούλια πλέον που έχουν συμφωνήσει να μην προσλαμβάνουν Εβραίους. Τέτοια έχουμε να αντιμετωπίσουμε κύριε πρέσβη. Τέτοια εχθρότητα κατά το Ισραήλ. Δηλαδή πολύ λίγες ελπίδες υπάρχουν να υπάρξει υποστήριξη σε αυτή τη συμφωνία η οποία έχει λογικές βάσεις. Είναι ρεαλιστική και έχετε δίκιο δεν θα έπρεπε να συνεχίσουν να χάνουν ευκαιρίες οι Παλαιστίνοι και όπως ε, κάποιος είπε κάποτε δεν χάνουν ποτέ ευκαιρία να χάσουν ευκαιρία εδώ και 70 χρόνια. Αλλά αυτός ο αντισημιτισμός που βλέπουμε παντού στην Ευρώπη είναι απειλή για όλους και απειλή για την Ευρώπη πάνω απ' όλα. Και φεύγουν από τις δυτικές χώρες της Ευρώπης οι Εβραίοι γι' αυτό το λόγο. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βελανουέβα εκ μέρου τη Γκουέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα καθυστερήσω ούτε ένα λεπτό να καταδικάσω τις βαρβαρότητες, τα απερίγρατα σχόλια των συμπολιτών μου εδώ, συνυπικών μου. Τέλος πάντων, ε, ε, πρώτα απ' όλα για να βρεθεί μια λύση πρέπει να έχει η Παλαιστινιακή Αρχή, το κράτος της Παλαιστίνης μια αξιοπρέπεια, χωρίς να έχει συνεχή εδαφική επικράτεια, χωρίς να μπορεί να διασυνδέσει τις περιοχές του με δρόμους, με ηλεκτρισμό, με νερό, κτλ. Την αποκάλεσαν συμφωνία του αιώνα. Πώς είναι δυνατόν να αποκαλούμε μια τέτοια, ένα τέτοιο σχέδιο, σχέδιο του αιώνα όταν το επεξεργάστηκαν χωρίς καθόλου να συμβουλευτούν την Παλαιστινιακή Αρχή. Η πρόταση αυτή είναι παράνομη πάνω απ' όλα. Και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξουμε το διεθνές δίκαιο. Και το διεθνές δίκαιο εδώ και Δεκαετίε προβλέπεται το διεθνέ δίκαιο και οι συμφωνίε των Ηνωμένων Εθνών την προστασία, την κοινή διαχείριση της Ιερουσαλήμ, να μην υπάρξει προσάρτηση στην κοιλάδα του Ιορδάνη, αφήνει στην κυβέρνηση την διαχείριση άνω των 10 εκατομμυρίων προσφύγων Παλαιστινίων στα εδάφη αυτά και τα αφήνει στη ζώνη του λικόφωτος. Δηλαδή θα συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν καθεστώ πρόσφυγα. Είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτή η συμφωνία ότι θα εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση, τα δικαιώματα ελεύθερης μετακίνησης. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε μια βιώσιμη ειρήνευση επί τη βάση ενό τέτοιου σχεδίου για τις επόμενες γενναίε. ποιε θα είναι οι συνέπειε, εάν ακούσουμε τι πιο εξτρεμιστικέ φωνέ τη χώρα σα για όλα αυτά. Ήδη ο ύπατος εκπρόσωπος ε, την περασμένη εβδομάδα ζήτησε να μην υπάρξει καμία μονομερής ε, κίνηση και πέραν του διεθνούς δικαίου υπάρχει και ο Γενικός Γραμματέας των ε, Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Γουτέρες, στις τελευταίες του δηλώσεις που αναφερθήκε στη ληστεία του αιώνα με την ευκαιρία αυτή. Και κύριε Πρέσβη, η, εάν η επιθυμία σας είναι η ειρήνη πρέπει να τηρήσετε το διεθνές δίκαιο. Πώς το Ισραήλ διατίθεται να συνεχίσει αυτή τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ. Thank you, colleagues. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Είναι πάντοτε από αυτά τα θέματα που είναι συναισθηματικά φορτισμένα. Το ξέρω. Παρ' όλα αυτά ας είμαστε κοινοβουλευτικοί εδώ στις, ε, στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμαστε. Ε, κύριε Πρέσβη, μία η ώρα πρέπει να τελειώσουμε τη συνάντησή μα τη συνέδριασή μα, γιατί στις 2.30 έχουμε ψηφοφορία. Δυστυχώ δεν μπορώ να πάρω άλλους να... να δώσουμε το λόγο σε άλλου αγορητέ. Θα δώσω το λόγο στον πρέσβη για 7-8 λεπτά για να συνοψίσει τη συζήτηση. Είστε σύμφωνο με αυτό? Ναι, απολύτως. Ε, και εγώ κάποια πράγματα θα τα έχω χάσει στη διερμηνία. Σας ε, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω στα ερωτήματα που τέθηκαν και εκφράζω βεβαίω και την εκτίμησή μου για το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται, για το διάλογο που έχουμε και θέλω να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι ο υπαριθμόν 1, 2 και 3 ε, ανησυχίες του Ισραήλ ε, είναι ανησυχίες ασφαλείας. Καθώς και ο υπαριθμόν ένα, δύο και τρία εχθρός της ασφάλειας του Ισραήλ είναι το Ιράν. Ξέρω φυσικά ότι όλοι έχουμε άποψη, είμαστε συναισθηματικά φορτισμένοι, αλλά πέραν όλων αυτών πρέπει να θυμάστε ότι το, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή που μιλούμε απειλείται από μια χώρα που για κάποιους από εσά είναι φίλη. Περιμένω από εσά λοιπόν ως ευρωβουλευτές και ως φίλοι του Ισραήλ που ενδιαφέρεστε για την ασφάλειά μας, όπως μόλις μου είπατε, να υψώσετε τη φωνή σας όταν το Ιράν απειλεί το Ισραήλ και όχι να παραμένετε σιωπηλοί. Δεν είναι συνεπές κάτι τέτοιο. Εμείς χρειαζόμαστε τη δική σας εμπιστοσύνη και εσείς χρειάζεστε τη δική μας εμπιστοσύνη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν αγνοείτε την υπαριθμόν ένα ανησυχία ασφαλείας του Ισραήλ. Δεν μπορεί να γίνει. Οπότε εμείς με χαρά να συνεχίσουμε τον διάλογο μαζί σας και με χαρά να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικές για εμάς αυτές, τις, ε, ε, ε, αυτές τις σχέσεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα. Όμως θα πρέπει ο ένας να αφουγκράζεται τον άλλον, όχι να εκτοξεύουμε εδώ πέρα αβάσιμες κατηγορίες. Τώρα, για το συγκεκριμένο ζήτημα της λύσης των δύο κρατών. Εγώ, ξέρετε, διπλωμάτης είμαι. Από αυτή την άποψη έχω την τύχη, χθες τη νύχτα, να έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργό μου σε τηλεοπτικό κανάλι Αραβο-Ισραηλινό. Και απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Ότι φυσικά και θα συζητηθεί αυτό το θέμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ποιο θα είναι λοιπόν ο στόχο των διαπραγματεύσεων, Να υπάρξει η, αυτή η διαπραγμάτευση. Εγώ δεν διαπραγματεύομαι, δεν διαπραγματεύομαι με τι αραβικέ χώρε του Αμερικάνους ή με τους Ευρωπαίους. Με τους Παλαιστίνιους πρέπει να διαπραγματευτούμε. μόλι συμφωνήσουν να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκεί πια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα πάντα, Συμπεριλαμβανόμενη και τη ενδεχόμενη λύση των δύο κρατών. Τέθηκε ένα ερώτημα για το Συμβούλιο ασφαλεία. Μα σε μένα το αποφθύνεται αυτό το ερώτημα. Δεν γίνεται. Εγώ εκπροσωπώ το κράτος του Ισραήλ. Ούτε τους Αμερικάνους, ούτε τους Ευρωπαίους, ούτε τους Άραβες, ούτε καν τους Παλαιστίνιους. Εγώ μιλώ εκ μέρους του κράτους του Ισραήλ. Αυτή είναι η χώρα μου. Και εμείς δεν είμαστε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ούτε έχει υπάρξει ποτέ μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας το Ισραήλ. Και αναρωτηθείτε κιόλα, για ποιο λόγο το Ισραήλ δεν έχει εκλεγεί ποτέ στο Συμβούλιο Ασφαλεία παρά τα 75 χρόνια ανεξαρτησία του. Γιατί η Ευρώπη δεν επιμένει το Ισραήλ να εκλεγεί μία φορά ω μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία. Δύο ευρωπαϊκέ χώρε μα έχουν προτείνει ω υποψήφια χώρα. Τη μία φορά που ε, υποβάλαμε υποψηφιότητα. Οπότε την, την αποσύραμε έναντι της Γερμανίας νομίζω και νομίζω η άλλη χώρα ήταν το Βέλγιο. Αλλά είναι και προς το δικό σας συμφέρον το Ισραήλ να μπει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Να μας υποστηρίξετε γιατί με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ θα αποκτήσει περισσότερη εμπιστοσύνη στο, στους διεθνείς οργανισμούς. Αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη μας είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δείτε τι έγινε στην, στην ε, Γενέβη. Έχουμε τη Βόρεια Κορέα και το Κατάρ και τη Βενεζουέλα να επικρίνουν το Ισραήλ. Αν είναι δυνατόν. Ε, πρέπει να είμαστε λίγο... Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Εγώ, ξέρετε, είμαι πολύ σοβαρό σε αυτό. Πρέπει να μα βοηθήσετε εσεί για να οικοδομηθεί περισσότερη εμπιστοσύνη από την πλευρά μα σε αυτού του ε, οργανισμού. Κύριε Μπάουζα, εκτιμώ αυτό που είπατε για τον, ασυ... για αντισημιτισμό. Φυσικά, βρίσκω αποτρόπαιο το φαινόμενο αυτό. Σε εσά εναπόκειται, εδώ σε αυτή την Επιτροπή, σε αυτό το Κοινοβούλιο, να καταπολεμήσετε ακόμη και εδώ μέσα τον αντισημιτισμό. Είναι ανησυχητική η έξαρση του αντισημιτισμού στην Ευρώπη. Το 2019 σημειώθηκαν τα περισσότερα αντισηματικά περιστατικά ε, από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ποιο είναι το μήνυμα που αποστέλλεται στους Ισραηλινούς πολίτες, στο κράτος του Ισραήλ, στους Εβραίους απανταχού της γης. Το αραβικό σχέδιο ειρήνευσης. Δεδομένου ότι οι Παλαιστίνοι έχουν δύο φορές απορρίψει ειρηνευτικά σχέδια τα οποία ήταν καλά για εκείνους, το 2008 ε, του Όλμερτ και το 2014 του Ομπάμα. Δεδομένου ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, οι πραγματικότητες έχουν αλλάξει και η Μέση Ανατολή είναι διαφορετική πλέον, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Πού είναι το σχέδιο Τραμπ. Αναγνωρίζω και αντιλαμβάνομαι ότι δεν θεωρούν όλοι αυτό το σχέδιο είναι καλό. Ε, ας επικεντρωθούμε στα θετικά αυτού του σχεδίου και ας διαπραγματευτούμε επί των όσων θεωρούμε ότι δεν είναι καλά στο σχέδιο αυτό. Κύρια Βιλανόβα, αναφερθήκατε στην Ιερουσαλήμ. Το 1947 το Ισραήλ, προτού καν γίνει κράτος, αποδέχθηκε τη λύση του διαχωρισμού. Ποιος αντιτάχθηκε τότε? όχι το Ισραήλ. Για 19 χρόνια μάλιστα οι Άγιοι Τόποι και η Ιερουσαλήμ βρίσκονταν υπό αραβικό έλεγχο και οι Εβραίοι δεν είχαν πρόσβαση στον ε, πιο ιερό τόπο του Ιουδαϊσμού για 19 χρόνια. Σήμερα το ίδιο αυτό σημείο είναι ανοιχτό προς όλες τις θρησκείες ακόμα και σε άτομα από χώρες με τις οποίες δεν έχουμε καν διπλωματικές σχέσεις. Ακόμα και από χώρες εχθρούς. Δίνουμε πρόσβαση σε ανθρώπους που έρχονται σε ανθρώπους προσκυνητές. Τους δίνουμε πρόσβαση στους Αγίους Τόπους. Αυτό είναι και ένας από τους λόγους που θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τον έλεγχο αυτών των Αγίων Τόπων. Γιατί έχουμε την, την εμπειρία, είναι αρνητική και δεν πρόκειται να την επιτρέψουμε να επαναληφθεί. Και τέλος, για τη δική σας ερώτηση και πάλι. Τι χρειάζεται το Ισραήλ για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Χρειαζόμαστε ένα Παλαιστίνιο εταίρο που θα έχει την προθυμία να έρθει και να διαπραγματευτεί μαζί μας. Αυτό και μόνο χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Και τους καλώ από αυτό το βήμα να το πράξουν. Να μην χάσουν για άλλη μια φορά την ευκαιρία. Γνωρίζουμε ότι δεν σας αρέσει το σχέδιο. Μπορεί να σας αρέσουν ελάχιστα σημεία του. Ελάτε όμως στο τραπέζι ε, διαπραγματευτείτε μαζί μας και στην πορεία μιας διαπραγμάτευσης πολλά μπορούν να συμβούν. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Συνάδελφοι, θα ξαναβρεθούμε εδώ στις ε, ψηφοφορίες, στις 2.30. Έχουμε την έκθεση για τη Λευκορωσία. Καλή όρεξη και καλό σας διάλειμμα.